Καλώ ήλθατε συνάδελφοι αυτήν την δεύτερη, στο δεύτερο τμήμα της συνεδριασής μας, όπου θα επικεντρωθούμε στο εθνικό και τοπικό επίπεδο. Έχουμε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων που θα μας εξηγήσουν τι κάνουν στα κοινοβούλια και τις αρμόδιες επιτροπές τους, όπως και εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και κοινωνική Επιτροπής. Όπως ήδη είδατε, έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία για μια εντελεχή συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και εκπροσώπων των κοινωνικών και οικονομικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωση. Όπως και στο πρώτο τμήμα της ε, συνάντηση. θα ζητήσω από τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που επιθυμούν να παρέμβουν, ε, στο τέλος ε, Τη συνεδρίαση να το κάνουν στο τέλος κάθε παρέμβασης, να χρησιμοποιήσουν τα ε, δελτία, τα ροζ που έχουν διανεμηθεί. Αλλά πριν από όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους συνεισηγητές της εκθέσεως της στρατηγικής εξέτασης ε, για την μετανάστευση. Η κυρία Ματσόλα δυστυχώς δεν είναι εδώ, αλλά ο κύριος Κοέλιο σίγουρα θα μπορέσει να σας ε, μεταφέρει κάποιες σκέψεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, αντικαθιστώ τον συνάδελφο Ρομπέρτο Μετσόλα που εκλήθη στην, ε, στις προπαρασκευαστικές εργασίες ε, τους, της σημερινής συνόδου. Μεταφέρω τα λόγια της συνοδευόμαστε εδώ μετά τη συμφωνία της ε, επανεγκατάστασης 160.000 ανθρώπων ή στην Ευρώπη μεταναστών διαδικασία που υπήρξε δύσκολη για αρκετά κράτη-μέλη και δυστυχώς απεκάλυψε ρογμές αντιθέσεις στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση Είμαι σίγουροι ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Πρόκειται για μια παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί μια παγκόσμια λύση με όλα τα κράτη και οργανισμούς εις το πεδίο. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρότυπο παράδειγμα σε αυτή τη διαδικασία. Εάν δεν υπάρξει μέλλον στις χώρες προέλευσης θα εξακολουθούν να προσέρχονται οι άνθρωποι αυτοί ανεξαρτήτως του κινδύνου για τη ζωή τους. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση αυτή προτού εξωθήσουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους ή στα χέρια των λαθρεμπόρων και διακινητών. Μόνον συνολικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και λύσεις με μέτρα μαζί με τις χώρες προέλευσης, διαμετακόμισης και προορισμού θα δώσει λύσεις. Και πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της ε, κοινή ε, εξωτερικής ε, πολιτικής και της μεταναστευτικής πολιτικής. Το μήνυμα αυτού εδώ του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να είναι ένα μήνυμα, ένα μήνυμα πολιτικών τσακωμών και διαφωνιών, αλλά ενότητας. Και γι' αυτό προετοιμάζεται μια έκθεση με συμμετοχή όλων των πολιτικών μερών, η οποία πρόκειται να απαντήσει ερωτήματα όπως η αλληλεγγύη και η δίκαιη κατανομή του βάρους της ευθύνης. Όπως και οι νομικές λύσεις για εκείνους που τη χρειάζονται, πού πηγαίνουν οι αεροαϊκοί πόροι ώστε να βοηθήσουν κάποιες χώρες να ξαναβρούν το δρόμο τους, πώς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης, πώς θα καταπολεμήσουμε τα δίκτυα διακίνησης, πώς μπορούν να προστατευτούν άνθρωποι πώς μπορούμε να έχουμε ένα πραγματικά κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και πώς μπορούμε να επιστρέψουμε εκείνους που δεν είναι επιλέξιμοι για καθεστώ προστασία στην Ευρώπη. Με την κατάσταση στη Συρία και την κρίση στη Λιβύη θα πρέπει να προετοιμάσουμε τα συστήματά μας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έρχονται και μάλιστα κατά μέτωπο, εξασφαλίζοντας ότι οι περιφερειακοί φορείς οι πόλεις, οι τοπικές αρχές θα έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν. Στο μεταξύ, η απάντηση δεν είναι να αμφισβητούμε το Σέγγεν ή τους εξωτερικούς συνοριακούς ελέγχους. Οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι περιορισμένοι και έχουμε καθήκον να τους χρησιμοποιούμε για εκείνους που περισσότερο τους έχουν ανάγκη. Όσοι δεν είναι επιλέξιμοι θα πρέπει να επιστραφούν. Ασφαλώς, αλλά ταχαίως. Πρέπει να βρούμε λύσεις και να συνεργαστούμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα συμβεί. Είμαι βέβαια ότι η σημερινή απογευματινή συνεδρίαση και οι συνεισφαρές σας θα είναι πολύτιμες και ελπίζω, υπολογίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να βρεθούν λύσεις. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο, λέει η Πρόεδρος. Κυρίε και κύριοι, περιμένουμε την κυρία Κέν και η οποία θα καταφτάσει από λεπτό σε λεπτό. Θα δώσω το λόγο στην Κέιτ Βάς, υπεύθυνο της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων ε, εκπροσωπώντας το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλώ. Ο κύριος Βάζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, μεγάλη τιμή για μένα που έρχομαι εδώ να μιλήσω εκ μέρου ε, της Δικής Επιτροπής της Βουλής των Κοινοτήτων για θέματα ε, εξωτερικών και συγχαίρω όλους για τη διοργάνωση της διάσκεψης. Χαίρομαι που κοινοβουλευτικοί συνάδελφοι William Cass, Stuart MacDonald και ο λόδος Τζέι είναι και αυτοί παρόντες και είναι προνόμιο για μένα να μιλώ στην αίθουσα Αναλίντ. Ήταν μία από τους μεγάλους κοινοβουλευτικού της Σουηδίας. Ήταν υπουργό ε, για θέματα ευρωπαϊκά στη χώρα της. Το πρόβλημα με τη μεταναστευτική κρίση και για το εκλογικό σώμα και τα εθνικά κοινοβούλια είναι πρόβλημα και το λέω σαν κάποιο που πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μοιράζεται τις αξίες της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε πάρα πολύ αργή στην αντιμετώπιση της ε, κρίσης και είδαμε φοβερές σκηνέ να εκτελήσονται, να περνάνε από χώρα σε χώρα μετανάστες, να τους προωθούν. Κάποιοι είχαν πληγεί από ε, αέριο, από τα κρυγόνα και είδαμε ότι ουσιαστικά προσπαθούν οι ηγέτες σήμερα που συνεδριάζουν να καλύψουν την υστέρηστη χρονική με αυτά που έπρεπε να γίνουν πριν και θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο και να μπορέσουμε να το πουλήσουμε στα εθνικά μας κοινοβούλια το σχέδιο αυτό και στο εκλογικό μας σώμα. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι στο κάτω-κάτω θα πρέπει να πούμε στον κόσμο που μας εκλέγει γιατί κάνουμε αυτά που κάνουμε. Δηλώνω ενδιαφέρον, είμαι μετανάστης στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πρόεδρος της Επιτροπής και εγώ πιθανότατα είμαστε οι μόνοι σε αυτή τη διάσκεψη που γεννήθηκαν στο Άντεν στην Ιεμένη. Ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν τριών ετών, εγώ όταν ήμουν εννέα. Έχουμε 40 ανθρώπους από εθνικές μειονότητες στη Βουλή των Κοινοτήτων και άλλους 40 στην Βουλή των Λόρδων. Οπότε συζητήσει αυτά τα θέματα που κατά το παρελθόν ήταν πολιτικής φύσεως τώρα είναι άκρος ευαίσθητα και απλά να συζητηθούν. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτά που θα κάνουμε στα κοινοβούλια μας θα τα εξηγούμε στους εκλογείς μας. Εγώ εκπροσωπώ την πόλη του Λέστερ, 60% του πληθυσμού του Λέστερ που ε, κατάγεται από την Ινδία, 20% από αυτούς είχαν απελαθεί ως πρόσφυγες από την ε, Αφρική. Και αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι τελικά να μην πηγαίνουν πιο γρήγορα από το εκλογικό μας σώμα όταν παίρνουμε αποφάσεις σε χώρους όπως αυτός. Θα πρέπει να περάσουμε σε μια περίοδο διπλωματίας δημόσια ανοιχτή για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι κάνουμε. Καλωσορίζω τα hot spots που έχουν δημιουργηθεί, αλλά έγιναν πολύ αργά. Πριν από δύο χρόνια η Επιτροπή μου πήγε στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας και εκεί είδαμε φρικτές σκηνές κόσμο προσπαθούσε να περάσει τα σύνορα. 100.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία τα έτη πριν το 2013 και η Ελλάδα και η Ιταλία εκλυπαρούσαν για βοήθεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις τώρα αποφάσισε να δώσει αυτή την υποστήριξη στις συζητήσεις μας στα Εθνικά Κοινοβούλια και σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια, αλλά όταν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των προσφύγων είναι κρίσιμη σημασία της χώρας και φοβάμαι ότι δεν βοηθούμε αρκετά την τουρκική κυβέρνηση όσον αφορά τους καταβλισμούς και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν και στο κάτω-κάτω ε, στο τέλος μένουν χωρίς την αναγκαία στήριξη θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή, να συνεχθούμε καλύτερα με τις χώρες Βορείου Αφρικής και θέλει η Επιτροπή μας να ξεκινήσει διάλογο με χώρες όπως είναι το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τινησία. Ε, δυστυχώς η κατάσταση στη Λιβύη είναι πολύ γνωστή. 92% του κόσμου που έφυγε από τη Βόρεια Αφρική και πήγε στην Ιταλία προερχόταν από τη Λιβύη. Διότι αφού τελειώσαμε την ευρωπαϊκή μας εκστρατεία στη Λιβύη δεν αφήσαμε ε, μία αλλά πέντε διαφορετικές κυβερνήσεις και σαν αποτέλεσμα αυτού ε, η πίεση αυτή προσέθεσε στην ε, κρίση τη μεταναστευτική. Θα πρέπει και το σχέδιο μετεγκατάστασης να εξηγηθεί πολύ προσεκτικά. Βέβαια, όταν διαρρέσει κανείς 120.000 ανθρώπους στις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε έχεις 4.200 ανθρώπους για κάθε χώρα. Και δεν θα συμβεί αυτό, διότι κάποιες χώρες απλώς δεν θα μπορέσουν να τους δεχθούν. Ο Πρωθυπουργό μα, ο Ντέιβιτ Κάμερον, δεσμεύτηκε να υποδεχτεί 20.000, αλλά άμεσα από του καταβλισμού τη Συρία. Οπότε έρχομαι στα δύο τελικά μου σημεία. Πρώτα απ' όλα, είναι μου σημασία ε, το έργο τη Ευρωπόλ. Θα πρέπει να δείξουμε στα εθνικά μα κοινοβούλια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπόλ κάνει ό,τι μπορεί την καλύτερη δυνατή δουλειά για να αντιμετωπίσει τα ε, εγκληματικά κυκλώματα και δεν το έχουμε ακούσει αυτό να αναφέρεται αρκετά στη διάσκεψη. Ε, δισεκατομμύρια ευρώ έχουν κερδίσει αυτά τα κυκλώματα λόγω της μεταστευτικής κρίσης και θα συνεχίσουν να κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα. Άκουσα με τα χαράς από την Ευρωπόλ που είπε ότι 27.000 ύποπτοι υπάρχουν. Αλλά οι εκλογείς μας θέλουν να δουν τους ενόχους όχι μόνο να συλλαμβάνονται, αλλά να καταδικάζονται, να φυλακίζονται και να κατάσχονται και οι περιουσίες τους, διότι εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη δυστυχία που οδήγησε αυτή η εκμετάλλευση σε τόσο πολύ κόσμο που ε, διακινδυνεύει τη ζωή του για να διασχίσει τη Μεσόγειο και τόσοι πολλοί άνθρωποι πέθαναν και πεθαίνουν. Τέλος θέλω να πω ότι η κατάσταση στη Συρία είναι αντικείμενο εκτεταμένων συζητήσεων. Κάποιες χώρες θέλουν να βομβαρδίσουν τη Συρία. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικότατοι όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική σε αυτές τις περιστάσεις, διότι αν δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί θα δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση Άρα θα πρέπει να σταθούμε λίγο, να προβληματιστούμε σοβαρά για τα όσα κάνουμε στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής. Δεν θέλουμε μια επανάληψη των σφαλμάτων μας που κάναμε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και στη Λιβύη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Βάς, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Κέγκε ήρθε. Σας δίνω το λόγο κυρία Κέγκε, Είναι η συγγήτρια της έκθεσης πρωτοβουλίας, στρατηγικής πρωτοβουλίας της ΛΥΜΠΕ για την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη μιας ε, γενικής, σφαιρικής, παγκόσμιας προσέγγισης όσον αφορά τη μετανάστευση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί είχαμε τη δυνατότητα να επισέθουμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά ε, τη δημιουργία των hotspot. Όπως ήλπιζα, οι παρεμβάσει των ομιλητών μας επέτρεψαν να διαλύσουμε διάφορα προβλήματα και αμφιβολίες. Στη συνεδρίαση την απογευματινή όμως θα αναλύσουμε το θέμα υπό το θέμα της διαχείρισης του μετασταυτικού φαινομένου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πριν ξεκινήσω την παρέμβασή μου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ελπίζω πραγματικά ότι αυτή η πρώτη ευκαιρία της συζητήσεως θα ενταχθεί στα πλαίσια διαθρωμένης και μόνιμης συζητήσεως ε, εγώ πρώτη αναγνωρίζω τη σημασία πολιτικού διαλόγου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την όρημη εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών αρχών για να βελτιώσουμε τις σχετικές προδιαγραφές για τις συνθήκες υποδοχής και τις διαδικασίες χορηγήσεως ασύλου και για να δημιουργήσουμε καλές πρακτικές σε θέματα ένταξης. Και αναφέρομαι όλος ιδιαίτερος στην κατάρτιση και στην παροχή βοηθείας. Μόνο μέσω μιας διαδρομής κοινής έχοντας πάντα υπόψη την προστασία εκείνων που ξεφεύγουν από τον πόλεμο, τη δίωξη και τη φτώχεια και ταυτόχρονα τα δικαιώματα των πολιτών, τις ανάγκες των πολιτών, τις προσδοκίες τους. Αν τα κάνουμε αυτά θα πετύχουμε αποτελέσματα λύσεις αποτελεσματικές για την υποδοχή και την ένταξη. Όπως γνωρίζετε το Κοινοβούλιο ξεκίνησε μια πολιτική διαδρομή με πρόθεση να επιφέρει μια αλλαγή όσον αφορά την ευρωπαϊκή προσέγγιση στο μεταναστευτικό φαινόμενο. Είμαι συνεισηγήτρια μαζί με τη συνάδελφο Ρομπέρτα Ματσόλα σε μια έκθεση πρωτοβουλία, στρατηγική έκθεση που αφορά τη Μεσόγειο και την ανάγκη μια ολιστική προσέγγιση στο μεταναστευτικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα ήθελα να διευκρινίσω δεν το διαχειρίζεται κανεί με συνθήματα ξενοφοβικά ή ακόμα χειρότερα με τείχου και φράγματα ε, και με δακρυγόνα το χειρίζεται κανείς αυτό επενδύοντας σε δράσεις συγκεκριμένες μέσης ε, και μακροπρόθεσμης δράσης ε, και κατεπήγοντα μέτρα για να ανταποκριθούμε στην καταστροφή την ανθρωπιστική και να έχουμε διαθρομές πολιτικές που εφαρμόζουμε ούτως ώστε να ελέγξουμε το φαινόμενο καταπολεμώντας τις βαθιές ρίζες του. Η προσέγγιση μας σε αυτή την πολιτική διαδρομή θα μας οδηγήσει να αντιμετωπίσουμε όλες τις πτυχές που με το φαινόμενο ανάμεσα σε αυτές τις ανθρωπιστικές υποχρεώσεις διάσωσης και προστασίας, τη διαφύλαξη των ετούντων άσυλων, την καταπολέμηση της διακίνησης και του εμπορίου των ανθρώπων, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τρίτων χωρών, επίσης και τις δημογραφικές προκλήσεις της Ευρώπης. Χρειάζεται ένα όραμα συνολικό που δεν θα είναι κατασταλτικό από τη φύση του, αλλά θα είναι πολιτικής και διπλωματικής φύσης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βαθιά αίτια της μετανάστευσης, εξυπηρετώντας, χρησιμοποιώντας το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές προσκήνιο, με πλήρη συμμετοχή όλων των φορέων, των θεσμών, των κρατών μελών, των διεθνών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών, των τρίτων χωρών. Ευχαριστώ και των προτέρων τους ομιλητές για τη συνεισφορά τους που θα, ε, που θα κάνουν σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τσέν Και τώρα θα μιλήσουν οι προσκεκλημένοι. Παρακαλώ να μιλήσετε για ένα δεκάλεπτο το πολύ, ούτω ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση. Πρώτη παρέμβαση. Ο κ. Φανσουά Ντεκώστε, πρόεδρος της Επιτροπής ΣΥΒΕΞ, της Επιτροπής των Περιφερειών και συγητής της νομοδοτήσεως για το θεματολόγιο το ευρωπαϊκό για τη μετανάστευση. Κύριε Ντεκώστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να σας μιλήσω. Έτσι μπορώ να εκφράσω την άποψη τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που πολύ συχνά είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την υποδοχή των μεταναστευτικών ροών. Όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα ηθαγενείας της Επιτροπής των Περιφερειών και η Επιτροπή των Περιφερειών μου ανέθεσε το καθήκον να συντάξω μια έκθεση όσον αφορά το ευρωπαϊκό θεματολόγιο της μεταναστεύσεως. Κατάγομαι από μια περιοχή, τον Όρπα Αντικαλή, όπου βρίσκεται στη Βόρεια Γαλλία απέναντι από την Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια περιοχή που τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια έγινε σύμβολο της ε, αποτυχίας της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά τη μετανάστευση. Και όταν λέω αποτυχία είναι ταυτόχρονα η, αποτοχή, η αποτυχία του να ξεβρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί το σύνορο μεταξύ δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και αν η μια χώρα ανήκει στο χώρο Σέγγεν ενώ η άλλη χώρα δεν ανήκει στο χώρο Σέγγεν αλλά και οι δύο χώρες είναι κράτη-μέλη της ίδιας ε, ένωσης που είναι πολιτική ε, και συνεχώς γίνεται πιο στενή. Είναι ένα σύμβολο επίσης της ε, αδυναμίας διαχείρισης της υποδοχής των μεταναστευτικών ροών και τέλος ε, θα έθετα την παρέμβασή μου σήμερα το απόγευμα σε ένα πλαίσιο που θα καλούσα πλαίσιο ε, κατεπήγων. Κατεπήγων διότι πρέπει να σας πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει επιλογή. Πολύ συχνά αντιμετωπίζει αυτή την ε, κατάσταση που ξεπερνά κατά πολύ τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκλεγόμενοι λοιπόν από τις περιστάσεις και από τη θέση που βρίσκεται υποδέχεται τους μετανάστες στην περιοχή της. Υπάρχει μια ταχύτατη αύξηση των μεταναστευτικών ροών, αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει η τοπική αυτοδίκηση και αλλάζει γρήγορα ε, και αλλάζει και η εθνικότητα των μεταναστών. Αυτό προσωπεύει βέβαια μια πολιτική δέσμευση και υποχρέωση από πλευράς τοπικής ε, αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα είναι και μια υποχρέωση οικονομική. Την περασμένη εβδομάδα με αρκετά μέλη της ομάδας ADLE, του Επιτροπής των Περιφερειών, πήγαμε στο Καλέ για να μιλήσουμε κοσόπους του Δήμου. Ε, το κόστος είναι 4-5 εκατομμύρια ευρώ ήταν η απάντηση που δεχτήκαμε σε ερώτησή μας όσον αφορά το κόστος της διαχείρισης ε, της υποδοχής των μεταναστών ε, για το καλέ. Πέρα από τους αριθμούς και τα στοιχεία, αυτό που ήταν σημαντικό και με εντυπωσίασε ήταν που είδα ότι αυτά τα στοιχεία δεν είχαν αξιολογηθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την πόλη του Καλέ. Ξέρουμε όμως αυτή, σε αυτή την πόλη οι κάτοικοι εδώ και αρκετά χρόνια έχουν υποστεί αυτό το πρόβλημα, ανταποκρίθηκαν με την καρδιά τους και τη γενοδορία τους και συνοδεύουν την υποδοχή των μεταναστών και δεν έγινε μια εκτίμηση του κόστους που αντιπροσωπεύει αυτό, αλλά δεν δίστασαν παρόλα αυτά να δαπανίσουν από το δικό τους προπολογισμό οι κάτοικοι για να μπορούν να τους υποδεχτούν και ε, να ανταποκριθούν και στις υποχρεώσεις τις πολιτικές και τις υποχρεώσεις ανθρώπινες που υποδέχονται ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από την δυστυχία. Μας είπαν ότι ε, υπήρχε αντίκτυπος εκπρόσωποι του Δήμου ε, ότι χρειάστηκε να βελτιωθεί η ασφάλεια των μεταφορικών μέσων μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας ε, οι οδηγοί πρέπει κάθε μέρα να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του εργαλείου που χρησιμοποιούν, των φορτηγών τους. Ε, και για έναν μεταφορέα είναι 150.000 ευρώ παραπάνω αυτό κοστίζει για να είναι σίγουρος οδηγός ότι θα αποφύγει να είναι εκείνος ο οποίος θα υποστεί τις ποινές και σε περίπτωση ε, ελέγχου αν διαπιστωθεί ότι ε, μετέφερε κάποιο μετανάστη στο φορτηγό του χωρίς να το προσέξει μπορεί να πληρώσει πρόστιμο 2.800 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά το μηνύο περιθώριο που έχει ε, σε κέρδος για το αναφορτηγό για τις μεταφορές. Είναι κατεπήγον το πρόβλημα διότι σήμερα η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται σε κάθε τοπική, σε κάθε περιοχή από τη μία πλευρά υπάρχει γενοδορία η οποία ε, οδηγεί σε μια ανακούφιση των, προβλημάτων των μεταναστών. Επίση υπάρχει από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλοί κάτοικοι που διαρωτώνται γιατί ε, αυτή η προσπάθεια ε, πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο από αυτούς γιατί δεν βοηθούνται περισσότερο και είναι ένα θέμα πολιτικό, είναι θέμα συνοχής που τίθεται για όλο και αυξανόμενο αριθμό τοπικών αυτοδιοικήσεων είτε όσον αφορά τα σημεία εισόδου στην ε, επικράτεια της κοινότητας ή διαμετακόμισης διότι όπως τα παρατηρήσατε ε, δεν βασίζομαι σε σημείο εισόδου τη μαρτυρία μου σε σημείο διέλευσης Έχω εμπειρία εισηγητού όχι μόνο της εκθέσεως που ετοιμάζω για την Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών του Δεκεμβρίου, αλλά και του γενικού εισηγητή μια εκθέσεως που συνέταξα τον περασμένο χρόνο κατόπιν αιτήματο τη Ιταλική Προεδρία και διαπιστώνω ότι σήμερα το ευρωπαϊκό σχέδιο διακινδυνεύει. Η συνοχή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, η συνοχή των Ευρωπαίων όλοι μαζί υλοποιούν ένα πολιτικό πρόγραμμα και ένα πολιτικό σχέδιο, αλλά σήμερα το θέμα της μετανάστευσης ε, διχάζει τους Ευρωπαίους. Διαιρεί Επίσης τους ανθρώπους και εντός της Επιτροπής των Περιφερειών, δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια δικηβεύματα. Είναι πρεμιέρα αυτή και είμαι μάρτυρας αυτής της ταχείας εξέλιξης. Όλο το ευρωπαϊκό σχέδιο και πρόγραμμα διακινδυνεύει κινδυνεύει και θα πρέπει να δώσουμε απάντηση και σε αυτό το ερώτημα, ώστε να σώσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η έκθεσή μου για μία ακόμη φορά θα κραυγάζει λέγοντας ότι είναι επίγον το, το πρόβλημα προς επίλυση. Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται βοήθεια, ε, ε, χρειάζεται χρηματοδότηση. Τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζουν νέα κονδύλια, αλλά θα πρέπει η χρηματοδότηση να είναι προσβάσιμη ταχύτερα από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ταχύτερα αυτό ίσως να σημαίνει και πιο άμεσα Γνωρίζω καλά ότι ε, τα περισσότερα χρήματα πρέπει να περάσουν μέσω των οργανισμών των κατών μελών. Αν προσθέσουμε όμως και τους ενδιάμεσους μεταξύ των προϋπολογισμών και της τοπικής αυτοδίκησης, τελικά στο τέλος η τοπική αυτοδίκηση είναι εκείνη που είναι στερημένη και περιμένει να φτάσουν τα χρήματα. Θα πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα. Ξέρουμε ότι η κατάσταση αυτή είναι εξαιρετική Μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούν και εξαιρετικέ έκτακτε διαδικασίε. Θα προσέθετα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση επίση χρειάζεται περισσότερε πληροφορίε, διότι είναι στην πρώτη γραμμή τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι το ίδιο να υποδέχεται κανεί μετανάστε που προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική ή από τη Συρία ή από το Ιράκ ή από την Ερυθρέα. Ε, χρειαζόμαστε να μπορούμε να προετοιμαστούμε κι εμείς για να υποδεχθούμε αυτούς τους διάφορους πολιτισμούς και νοτροπίες Ξέρουμε ότι η γεωπολιτική έχει αναστατώσει πολλές χώρες που είναι γειτονικέ της Ευρώπης. Ξέρουμε όμως ότι και οι μετανάστες δεν είναι οι ίδιοι σήμερα και σε δέκα, δεν θα είναι οι ίδιοι σε δέκα μήνες. Άρα χρειαζόμαστε να μπορούμε να ενημερώνουμε τις τοπικές αρχές ώστε να μπορούν και αυτές να προβλέπουν το είδος της υποδοχής που απαιτείται και ούτως ή άλλως θα διοργανώσουν την υποδοχή για αυτούς τους μετανάστες. Βέβαια, ε, πέρσι και φέτος βασική λέξη της εκθεσής μου είναι η αλληλεγγύη. Ε, μια αλληλεγγύη που ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε επίσης να στηρίξει την όλη προσπάθεια της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 80. Ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να συζητάμε πλέον μεταξύ μας τα, θα πρέπει κατεπηγόντως να ανταποκριθούμε, να βρούμε απάντηση ξεκινώντας ε, από το άρθρο αυτό που εγκαθιδρεί την αλληλεγγύη όχι μεταξύ των κρατών μελών και μόνο και γι' αυτό είμαι και εδώ σήμερα αλλά και προς την τοπική αυτοδιοίκηση, τις τοπικές αρχές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ε, τον κύριο Κιώστερ. Η μεγάλη πλειοψηφία των θεμάτων αυτών τίθενται για όλους και πρέπει να βρούμε απαντήσεις όλοι μαζί τα ερωτήματα αυτά είναι αλήθεια. Θα συνεχίσουμε τώρα με του εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λαμάριο, ε, πρόεδρος της Κοινοβουλικής Επιτροπής Ιστορικών Θεμάτων από την Κύπρο. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Αυτό το Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, για χρόνια τονίζαμε σε ανάλογες συναντήσεις και στη ΚΟΣΑΚ πλήστες φορές την ανάγκη συλλογικής ενασχόλησης με το θέμα της μετανάστευσης με τρόπο σφαιρικό και σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για χρόνια προσπαθούσαμε να ευαισθητοποιήσουμε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πίεση που δεχόμασταν ως χώρες της Μεσογείου από τις μεταναστευτικές ροές. Δυστυχώς χρειάστηκε να υπάρξουν κατ' επανάληψη άνευ προηγουμένου ανθρώπινες τραγωδίες στη Μεσόγειο με θύματα ακόμη και αθώα παιδιά. Η πρόσφατη δε του διαδρόμου σε εισαγωγικά των Δυτικών Βαλκανίων ανάγκασε περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δουν το μέγεθος του προβλήματος και να αναζητήσουν μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο θέμα. Αυτό βέβαια είναι και ενδεικτικό του τρόπου λειτουργίας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αντιδρούμε αντί να δρούμε προληπτικά, δίνοντας πρόσκαιρες λύσεις με μηδενικά ή τουλάχιστον ασήμαντα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές. Είναι όμως η αποσπασματική αντιμετώπιση στην προσφυγική κρίση όπως την ονομάσαμε τρόπος αντίδρασης. Είναι η διοχέτευση των προσφύγων στις παραδίπλα χώρες ή πολύ περισσότερο το κλείσιμο των συνόρων λύση. Για εμάς είναι ξεκάθαρο και το υπογραμμίζουμε ξανά. Το θέμα της μετανάστευσης θα βρίσκεται μπροστά μας όσο οι συγκρούσεις στις γύρω περιοχές και η έκρηθμη κατάσταση συνεχίζονται. Επομένως, Κύριε, πρέπει να εργαστούμε για την καταπολέμηση των βασικών αιτιών της μετανάστευσης και πρώτιστα τις πολεμικές συγκρούσεις που επιτείνουν τη φτώχεια, την έλλειψη δημοκρατίας και την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, ορισμένες επιλογές και η ανικανότητα να δράσουμε αποτελεσματικά δεν συνέβαλαν στο να δημιουργηθούν συνθήκες ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης στις χώρες της άμεσης γειτονίας αλλά και στη γειτονιά των γειτόνων μας από όπου προέρχονται κύρια τα μεταναστευτικά ρεύματα. Καταλητικό στοιχείο αποτελεί διαχρονική πολιτική ορισμένων ισχυρών οικονομικά χωρών που ευθύνονται για την εκμετάλλευση άλλων χωρών με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανισορροπιών στο εσωτερικό του και την άνθηση μη δημοκρατικών καθεστώτων. Μακάρι η αυτοκριτική μερικών ηγετών στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρώπη που θέλουν να ζουν, αλλά και την κριτική του κύριου Γιούγκερ για πολιτικές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οδηγήσουν σε αίσια ανέκβαση διεργασιών για ολιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος. Ανησυχούμε ότι η έλλειψη της απαιτούμενη πολιτικής βούλησης μπορεί να οδηγήσει σε ημίμετρα τα οποία αντί να συμβάλλουν στην προσωρινή τουλάχιστον άμβληση του προβλήματος θα επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες αφού πολλές πτυχές του ζητήματος δεν θα τύχουν επαρκούς αντιμετώπισης. Θεωρούμε πως πρέπει να είναι πλέον ξεκάθαρο στον καθένα μέσα και από τα πρόσφατα γεγονότα τι καθημερινά μεταναστευτικές ροές και την προσφυγική κρίση πως αυτά δεν αφορούν μόνο ένα κράτος ή μόνο μια ομάδα κρατών αλλά επηρεάζουν το σύνολο της Ένωσης. Η όποια επομένως ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση θα πρέπει να εκπονείται τοποθετώντα στο επίκεντρο του πνεύματος των αποφάσεων την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Σε αυτά τα πλαίσια, μέσα από κοινή συμφωνία και δράση, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί και το θέμα της μετεγκατάστασης των προσφύγων. Έχει μια ξεχωριστή σημασία, δεδομένου ότι το θέμα της μετανάστευσης δεν αναμένεται να αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά, ούτε να απαλληφθεί διαπαντός λόγω των βαθύτερων αιτιών που αναφέρθηκα προηγουμένω. Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα του θέματος, συζήτησε διεξοδικά σε επίπεδο ολομέλειας του σώματος θέμα με τίτλο «Τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στην Μεσόγειο». Στα πλαίσια αυτά κάλεσε τον περασμένο Μάη τον αρμόδιο επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Αβραμόπουλο, και ενημέρωσε το Σώμα για την πολιτική τη Ένωση στον τομέα της μετανάστευσης. Σε δεύτερη συνεδρία η Ολομέλεια του Σώματος ήγηρε σειρά πτυχών του ζητήματος που αντικατοπτρίζουν πολύ και τα όσα προανάφερα. Ασκήθηκε κριτική για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεντρώθηκε η συζήτηση κυρίως στην αντιμετώπιση προβλημάτων των χωρών προέλευσης των προσφύγων με επίκεντρο τη δημιουργία συχτικών ευημερία, ασφάλεια, ειρήνη και ανάπτυξη, ώστε να υπάρξει μακροπρόθεσμο και ουσιαστικό αποτέλεσμα σημειώθηκε η ανάγκη άμεση εφαρμογή τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, η οποία να στηρίζεται στι αρχέ αλληλεγγύη και τη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και στο σεβασμό τη αξία τη ζωή. Συναφώ εκφράστηκε και η άποψη υπέρ τη άμεση αλλαγή του κανονισμού Δουβλίνο 2. Αφού εκτιμήθηκε το έργο του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας προτάθηκαν μέτρα προστασίας από τα δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών και τα τυχόν τοπικά κυκλώματα δουλεμπορίου που δρούσε σε κάποιες χώρες. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη λήψης πιο αποτελεσματικών μέτρων για καταπολέμηση της παράνομης εργασίας και της εργασιακής εκμετάλλευσης των μεταναστών. Τονίστηκε ακόμη η ανάγκη αντιμετώπισης των προσφύγων και νόμιμων μεταναστών. Ακόμη, η, η βάση των διεθνών και ευρωπαϊκών κανόνων και προτύπων, καθώς και οι ανάγκες σωμάτωσης στις τοπικές κοινωνίες, ενημέρωσης τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, αλλά και την εκπόνηση πολιτικής ενάντια στο ρατσισμό. Υπήρξε συζήτηση για τα προβλήματα της οικογενειακής επανένωσης ή της έκδοσης αδειών παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Με αυτά τα ζητήματα ασχολήθηκε επίσης η Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όπως και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών. Για τη χώρα μας, συνάδελφοι, η σημασία που προσδίδουμε στο θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου έχει μια άλλη διάσταση συνδεδεμένη με την ιδιότητα του πρόσφυγα που χαρακτηρίζει πολλούς από τους συμπατριώτες μας Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους από τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974. Είναι για μα και για αυτόν τον λόγο μίζο θέμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η αλληλεγγύη υπέρ όλων των ατόμων που διαφεύγουν από συγκρούσεις, διωγμούς, την αστάθεια και τη φτώχεια στη χώρα τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φίλου ή θρησκείας. Η Κύπρος, βάσει της πρότασης που συζητήθηκε στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών στις 14 Σεπτεμβρίου, θα δεχτεί ευχαρίστως την μετεγκατάσταση στο έδαφο τη. 274 προσφύγων από την Ουγγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία, με αποτέλεσμα να ανέλθει ο αριθμό των ατόμων με το καθεστώ πολιτικού πρόσφυγα πέραν των 500. Εξαιρουμένων των όσων έχουμε εμεί στη χώρα μα σε κέντρα υποδοχή, οι οποίοι πρέπει να εγκατασταθούν αλλού γιατί ήδη το θέλουν. Δεδομένου ότι ο πληθυσμό τη Κύπρου είναι μικρότερο του ενό εκατομμυρίου και υπό το φω τη οικονομική κρίση και ψηλή ανεργία που μα ζητήσουν τη χώρα μα, ο αριθμός αυτός είναι σημαντικός. Ακόμη το πρόβλημα επιτείνεται και από την παράνομη είσοδο μεταναστών από το γεγονός ότι η νόμιμη κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου με αποτέλεσμα από την γραμμή αντιπαράδεξη να μπορούν να εισέλθουν παράνομα αρκετοί προερχόμενοι από την Τουρκία. Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλώντα για τη μεταναστευτική πολιτική, πρέπει να έχουμε συνεχώ κατά νου ότι πρόκειται για μια πολιτική που φορά ανθρώπου. Πρόκειται για θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας που πρέπει να διασφαλιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λάμαρη. Ο κύριος Μιλιόρε, πρόεδρος της Επιτροπής Ερεύνης ε, για την υποδοχή, ταυτοποίηση και κράτηση των μεταναστών από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσω Πρόεδρε, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για αυτήν την πολύ σημαντική διακοινοβουλευτική συνεδρίαση εμείς είμαστε περήφανοι που μπορούμε να εκπροσωπούμε θα εδώ μαζί με τη συνάδελφο Σεντέμερο και τους υπόλοι... τα υπόλοιπα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας και τους υπόλοιπους ε, συνεισηγητές ώστε να τοποθετηθούμε σχετικά με τις κατευθύνσεις που η χώρα μας επιθυμεί να ακολουθηθούν σε αυτό το πεδίο που είναι όλο και πιο κρίσιμο. Κρίσιμο ακόμα και για την ίδια την ε, ουσία της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση αυτή όταν μιλούμε για ολιστική προσέγγιση εννοούμε ότι δεν θέλουμε περιοριστικές προσεγγίσεις. Ότι δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε όλες τις πτυχές, τις πτυχές και τα επίπεδα του προβλήματος και να τις βλέπουμε με το πιο διαθρωμένο τρόπο. Ιδάλλως θα έχουμε τα ίδια λάθη ε, σαν να ήθελε κανείς να εξετάσει το φαινόμενο της ζωής και να το εξέταζε μόνο χημικά ή βιολογικά, λέει ο Όλες αυτές λοιπόν οι, τα κρούσματα, οι περιπτώσεις ε, κρίσεως, τραγωδίας ανθρώπινης που διέπουν αυτές τις ροές, χωρίς να μιλούμε για τον περιορισμό τους, σαν ξαφνικά να παρέκυψαν ενεθρία βέβαια αυτές οι ροές, και διατηρώντας αυτήν την ολιστική, όπως λέμε, προσέγγιση, έχουμε ένα σημαντικό στοιχείο εδώ, τη συλλογική μνήμη που συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, την Μεσόγειο και την Ιταλία που ήταν πάντοτε πατρίδα προσφύγων που διέφευγαν από απολυταρχικά καθεστώτα, από πολέμους, από σειράξεις. Εδώ μιλούμε για ένα από τα πιο θεμελιώδη στοιχεία για να καταλάβουμε το ρόλο που διαδραματίζουμε εδώ και την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού αυτού οράματος και σχεδίου αλλά και τις θεμελιακές αρχές αυτές της εβραϊκής μας Ένωσης που την ιδρύσαμε για να ξεπεράσουμε τους πολέμους, να γκρεμίσουμε τους τείχους και να μην τους ξαναχτίσουμε ποτέ. Το κοινωνικό, το πολιτιακό, οικονομικό πρότυπο δεν αμφισβητείται από τους μετανάστες ή στην Ευρώπη, αλλά από αυτούς που αρνούνται τις αξίες μας στην Ευρώπη. Τα στοιχεία δηλαδή, τα ιδιαίτερα στοιχεία του πολιτισμού μας. Το δικαίωμα στο άσυλο είναι θεμελιώδες και ατομικό. Και για τον λόγο αυτόν θεωρώ ότι η περίπτωση στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μορκόνε, δηλαδή το ευαίσθητο του ζητήματος, σχετικά με το να καταρτήσουμε κατάλογο ασφαλών χωρών, ώστε να ταυτοποιήσουμε αυτούς που ζητούν διεθνή προστασία ή άσυλο, πρέπει να το βλέπουμε υπό την έννοια της εγγύησης των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και είναι δικαίωμα όλων, όλων μας. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό είναι θεμελιώδης και η προσπάθεια που καταβάλει η χώρα μας να προωθηθεί μια πολιτική ενίσχυσης όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών της ΕΑΣΟ και των υπολείπων που διέπουν τα ανθρωπιστικά στοιχεία της μετανάστευσης και την αποτελεσματικότητα του, της διαδικασίας επαναπατρισμού πάντοτε με την προστασία των θεμελιωδών και ανθρώπινων δικαιωμάτων και στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Δουβλίνου. Για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι είναι πραγματικά ουσιαστικότατο να επικαιροποιήσουμε και την εθνική μας νομοθεσία σχετικά με τις νόμιμες διόδους και των προσφύγων δηλαδή τη δυνατότητά τους να προσέρχονται απευθείας σε ε, εγκαταστάσεις διαμετακόμισης και θέλοντας να αντιμετωπίσουμε την υποκρισία τα τελευταία 20 χρόνια από 500.000 περάσαμε σε 5,5 εκατομμύρια οι περισσότεροι παράνομοι και σιγά σιγά νομιμοποιούμενοι με μεταβατικές και έκτακτες διαδικασίες συνεχώς. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να προωθήσουμε προς τα εμπρός ένα ενιαίο πρότυπο υποδοχής και ασύλου πανευρωπαϊκό και μια εντατικοποίηση των ελέγχων. Γιατί από τη στιγμή που το δική, δικό μας σύστημα ασύλου είχε κενά και ελλείψεις δεν το κρύψαμε. Το θέσαμε σε μια επιτροπή ερεύνης που ως πρώτο πόρισμα η επιτροπή μας είχε το εξής και λέω κάτι κοινότυπο αλλά αυτές οι ροές είναι που μπορούν να οδηγήσουν πιο εύκολα σε εγκληματικές τάσεις και εγκληματική δραστηριότητα και εσωτερικά και εξωτερικά. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι αυτοί που υποδεχόμαστε είναι άνθρωποι με τραυματικές αμπειρίες και στη διαμετακόμιση τους και ακόμα και στην παραμονή τους. Δεν μιλούμε απλώς για διακινητές και λαθρεμπόρους που πραγματοποιούν παράνομα κέρδη. Πολύ συχνά είναι και ε, σαδιστικής φύσεως ε, τύρανοι αν θέλετε. Επομένως πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης και συνεχούς ενημέρωσης όλων των αρμοδίων από τους αστυνομικούς μέχρι τους υγειονομικούς, από τους διοικητικούς μέχρι την ίδια την κατηγορία των πολιτικών ηθινόντων. Και επίσης ένα επιχείρημα που δεν εθίχθη στο βήμα αυτό, αλλά που έχω την εντύπωση ότι είναι θεμελιώδης για να δώσει και αξιοπιστία στην πολιτική μας πρωτοβουλία, δηλαδή εκείνο της ενημέρωσης γνωρίζουμε πόσο είναι απαραίτητο να έχουμε σωστή και πλήρη ενημέρωση, διότι η αγορά του τρόμου, η πολιτική αγορά του φόβου και του τρόμου εκμεταλλεύεται τις ε, προκατασκευασμένες εικόνες ε, που αποκλίνουν από την πραγματικότητα. Πρέπει να εστιαστούμε στο παιδαγωγικό και σχολικό πρόγραμμα, στα μέσα ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται μια ισορροπημένη και σωστή ενημέρωση σχετικά με την πραγματικότητα. Η με αφορά αυτό είναι απολύτως θεμελιώδες. Κατά τα άλλα, παρά την προσοχή που έχει δοθεί στη χώρα μας σε κάποια φαινόμενα διαμαρτυρίας σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας σχετικά με την προσέλευση μεταναστών ή προσφύγων, αυτά είναι μειονοτικές τάσεις στη χώρα μας, οι οποίες όμως κάνουν πολύ φασαρία και μέσω των μέσων ακριβώς ενημέρωσης πολλαπλασιάζεται η φωνή τους και φαίνεται ότι είναι πιο μεγάλες τάσεις από αυτό που στην πραγματικότητα είναι. Πρέπει λοιπόν να εισαγάγουμε στοιχεία εξορθολογισμού και να βλέπουμε ε, την ανθρωπιστική μας προσπάθεια πάντοτε σε ένα πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πέρασμα και ρισκάρει πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια τη στην και το λέγω αυτό ως εκπρόσωπος Εθνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός. Θα πρέπει, θα πρέπει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπους να αναλάβουμε. Γιατί αλλιώς αν δεν μπορούμε αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδων να αναλάβουμε, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα 500 εκατομμύρια των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ κύριε Μιλιόρα. Ο κύριος Μάρκεθ Ντελαρούβια από την Επιτροπή Ιστορικών Θεμάτων από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Καλησπέρα Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφραστώ σήμερα στα Ισπανικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει εγγράψει και έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα εθνικά συντάγματα και από τις διατάξεις των νομοθεσιών των κρατών μελών. Υποτείνει αυτή όλες οι πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στην πολιτική μετανάστευση, όπως και για τις υπόλοιπες πολιτικές, βασίζονται στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων η οποία αναγνωράζει, θυμίζουμε, κάποια άλλα δικαιώματα όπως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ελευθερία, στην ασφάλεια, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, ελευθερία εργασίας και το δικαίωμα του ασύλου. Σε περίπτωση ε, ε έκδοσης από κάποια χώρα ε, και το δικαίωμα στη μη διακριτική μεταχείριση. Επομένως δεν είναι μόνο οι διατάξεις που αφορούν στα εθνικά συντάγματα. Αυτά έχουν εγγραφεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο σε επίπεδο συνθήκη, σε επίπεδο δηλαδή χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τώρα μέσω της ε, τραγωδίας που παρακολουθούμε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αυτή τη στιγμή συζητούν την δυνατότητα ανάληψης νέων μέτρων σε μια ευρύτατη εστίαση στα θέματα μετανάστευσης. Επομένως θεωρώ ότι η πρόσκληση σε αυτήν τη συνεδρίαση δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Πραγματικά αντιμετωπίζομαι μια έκτακτη ανάγκη και οι έκτακτες ανάγκες χρειάζονται άμεση ανταπόκριση και χρειάζονται άμεσα βραχυπρόθεσμα και χρειάζονται ευφυή διαχείριση μακροπρόθεσμα. Η Ισπανία καταβάλει ήδη την προσπάθεια δημοσιονομική για να διατηρήσει προγράμματα υποδοχής ετούντων ε, άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας και επομένως αυτές οι χρηματοδοτήσεις δεν έχουν υποστεί καμία μείωση στα τελευταία, στους τελευταίους προϋπολογισμούς που εγκρίναμε, κάθε άλλο αυξήθηκαν ελαφρά σε αντίθεση με τους εβραϊκούς πόρους που αφιερώνονται στις προσπάθειες αυτές. Και θυμίζω σε χώρα η οποία ε, περνάει από πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια. Καμία χώρα από αυτές που είναι γύρω μας δεν προσφέρει τόσο πολυετή και μακροπρόθεσμα προγράμματα, προγράμματα υποδοχής και ένταξης κοινωνικής όπως και εργασιακής και αυτό το κάνουμε αποφασισμένα, αλλά το κάνουμε και υπεύθυνα ανάλογα με τις δυνατότητες υποδοχής μας. Που στην Ισπανία υπολογίζεται απέναντι στην ευθύνη που έχουμε στους χιλιάδες ανθρώπους που προσέρχονται στο έδαφος μας και για οικονομικούς λόγους. Γίνεται αυτό μέσω κέντρων και υπηρεσιών συγκεκριμένων των Υπουργείων, των Αρμοδίων, αλλά και μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν εξειδικευτεί στο πεδίο αυτό. Υπό την έννοια αυτή, η Ισπανική κυβέρνηση ήδη ενέκρινε τα πρώτα στοιχεία στα πλαίσια της συμφωνίας του σχεδίου Juncker της ε, επανεγκατάστασης και είμαστε έτοιμοι ε, στο πλαίσιο της συμφωνίας που τελικά θα εγκριθεί είτε ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είτε στα πλαίσια επιμέρους συμφωνιών τις ποσοστώσεις που θα μας αλλαγωνούν. Η εγκύτητά μας στην Αφρικανική Ήπειρο και τα εκατοντάδες χιλιάδων ε, χιλιόμετρα εξωτερικών συνόρων που έχουμε μας αποκαλύπτουν σε τεράστια πίεση. Το 2006 προσήλθαν δεκάδες χιλιάδων, έκτοτε αυτές οι ροές έχουν συνεχώς ε, ενταθεί οδηγώντας σε ε, ανθρωπιστικές κρίσεις και στις επανειλημμένες, ε, στα επανειλημμένα επεισόδια ε, των, εγκληματικών δραστηριοτήτων διακινητών και λαθρυμπόρων. Από το 2006 ως σήμερα έχει αυξηθεί κατά 90 και πλέον της 100 η προσέλευση παράνομων μεταναστών στα εδαφών μας. θα πρέπει όλες οι χώρες μαζί να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε ή να διαχειριστούμε καλύτερα τις ροές αυτές μέσω και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εξωτερική Διαχείριση των ε, Συνόρων, της Frontex δηλαδή, όπως και άλλων φορέων και οργανισμών που εργάζονται στο πεδίο αυτό. Ως πρότυπο της συνεργασίας αυτής, εγώ θα ήθελα να αναφέρω τη στενή συνεργασία που έχουμε με το Μαρόκο, τη Σενεγάλη ή τη Μαυριτανία, χάρη στη συνεργασία με τις οποίες τουλάχιστον στις Κανάριες ε, μίσους είχαμε σημαντική μείωση της παράνομης μετανάστευσης. Θα ήθελα τώρα να υποκαναμίσω κάποια πράγματα. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι η μετανάστευση είναι η σημαντική και μεγάλη πρόκληση εποχής μας. Είναι και θα είναι. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε η, η Ευρώπη να μεταμορφωθεί σε ένα οχυρωμένο φρούριο κάστρο. Πρέπει να διατηρήσουμε τις αρχές αλληλεγγύης μας Επομένως δεν πρόκειται ούτε για εξωτερικά σύνορα ούτε για φράχτες, αλλά για διαχείριση των πόρων μας, των δυνατοτήτων μας και όλων των κοινωνικών φορέων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πεδίο αυτό. Το κλειδί βρίσκεται στο να κατανοήσουμε ότι η βελτίωση των συνδικών ζωής στις χώρες προελεύσεως είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στο πλαίσιο του δράματος αυτού. Μία αποτελεσματική συνεργασία με τι χώρες αυτής προέλευση είναι ο μόνος τρόπος μέσω της βελτίωση των συνθηκών ζωή των πολιτών τους να επιλύσουμε το πρόβλημα ε, με, αποτελεσματικό και ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο τρόπο. Η αλληλεγγύη βεβαίω είναι ο μεγάλος πυλώνας της ε, ενώσης των πολιτισμένων χωρών αλλά και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, γιατί αυτή είναι μια προσπάθεια που θα πρέπει να μοιράζεται το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. μέσω των φορέων της και των οργανισμών της. Χρειάζεται στήριξη οικονομική και πολιτική και διοικητική για τις χώρες αυτές που υφίστανται τη μεγαλύτερη πίεση στα εξωτερικά του σύνορα. Και η στήριξη αυτή θα πρέπει να δίδεται και στις τρίτες χώρες που είναι χώρες προέλευσης ή διαμετακόμισης των προσφύγων και των μεταναστών. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, αποτελεσματικούς μηχανισμούς συνεργασίας με τις χώρες αυτές μέσω και μακροπρόθεσμα. Χρειάζεται επίσης μια κοινή διαδικασία και κοινή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που να στηρίζεται στην ιστορική μας δυνατότητα να προσφέρουμε συνθήκες διαβίωσης και υποδοχής και στην καταπολέμηση των, οργανωμένων εγκληματικών οργανώσεων διακινητών. Η παράνομη μετανάστευση είναι το πεδίο στο οποίο άνθρωποι γίνονται θύματα εκμετάλλευσης, αυτό, αυτά τα φαινόμενα αυξάνονται εντυπωσιακά και επομένως είναι υπαριθμόν ένα προτεραιότητά μας να το καταπολεμήσουμε. Εμείς έχουμε ζήσει από πολύ κοντά τα προβλήματα αυτά και θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποιες ε, λύσεις ή κατευθύνσεις προς λύσεις. Όλοι έχουμε κάνει επίσης λάθες. Όταν προσφέρουμε εύκολες λύσεις στους, ε, στην παράνομη διαβίωση των ε, μεταναστών δεν κάνουμε παρά να διευκολύνουμε το έργο των διακινητών και των λαθρεμπόρων. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε κατεπηγόντως τις συμφωνίες του Δουβλίνου που έχουν μετατραπεί σε κενό γράμμα αυτή τη στιγμή. Και ελέγχθηκε σήμερα. Πρέπει να ξαναδούμε τα μέσα που έχει στη διαθεσή της η Frontex. Θα πρέπει με αποφασιστικό τρόπο να ξαναεξετάσουμε τα, τα διαβόητα hot spot που είναι αντικείμενο συζήτησης όλες αυτές τις μέρες και βεβαίως σήμερα. Και θα πρέπει να πάμε σε ταχύτατη επιστροφή όλων εκείνων των ανθρώπων που δεν είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ή ασύλου. Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια, αλλά όπως το είναι και οι κίνδυνοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Ντελαρουμπία. Σίγουρα έχετε μεγάλη εμπειρία στον τομέα της μετανάστευσης. Φίξατε ένα σημαντικότατο ζήτημα το οποίο ελπίζω να είναι το επόμενο στάδιο. Δηλαδή τα προγράμματα ένταξης όλων αυτών που έρχονται στην Ευρώπη και ήρθαν στην Ευρώπη. Να δώσω το λόγο στην κυρία Κάρι Χάριξεν της Επιτροπής δικαιοσύνη του Νορβηγικού Κοινοβουλίου. Η Νορβηγία δεν είναι μέλλον της Ένωσης, συμμετέχει ε, στο... Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρέμβαση και είναι πολύ ενδιαφέρουσα για μας, για την Ένωση, να ξέρουμε ε, ποια είναι η άποψη της χώρας. Η κυρία Άνριξεν, λοιπόν, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε να έρθω εδώ. Είναι ιδιαίτερα σε αυτές οι συζητήσεις τα άλλα εθνικά κοινοβούλια για εμάς, για αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει τόσο τραγικές ε, επιπτώσεις. Αυτή η κρίση είναι η αρχή μιας κρίσης για όλη την Ευρώπη. Είναι αδύνατο να επιστρέψουμε στην κατάσταση που βρισκόμασταν πριν την αρχή της ε, κρίσης. Είναι μια κρίση που θα μας οδηγήσει σε κάτι τελείως ε, καινούριο και διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν η Νορβηγία στηρίζει και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ολιστικές προσεγγίσεις για δημοκρατική και ειρηνική ε, εξέλιξη στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες. Η κρίση... Η μεταναστευτική κρίση είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντική για την Νορβηγία και ήταν και ένα θέμα στις πρόσφατες εκλογές που είχαμε. Ο πληθυσμός της ε, Νορβηγίας, οι πολίτες της Νορβηγίας θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτήν την προσπάθεια. Και θα ήθελα να προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί είναι αυτή η κρίση κάτι που αφορά και εμάς και να σας ενημερώσω για τα κύρια στοιχεία μιας πολιτικής συμφωνίας που ολοκληρώθηκε στο Κοινοβούλιο μας πριν ε, το καλοκαίρι. Και τέλος θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένες, ε, ορισμένα στοιχεία που προσφέρει η Νορβηγία σε αυτήν την αντιμετώπιση. Καταρχάς, η Νορβηγία συμμετέχει σε πάρα πολλά ε, κομμάτια της συνεργασίας στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, είναι μέλος του Σέγγεν, της συνεργασίας του Δουβλίνου και του Ευρωπαϊκού ε, Γραφείου για ε, το Άσυλο και ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στον αριθμό των ετούντων άσυλων στην Νορβηγία. Οι αριθμοί από το Γραφείο Μετανάστευσης της Νορβηγίας ε, για το 2014 δείχνουν πως 11.500 ετούτες άσυλο έφτασαν στην Νορβηγία. Εκτιμάται ότι οι αιτήσει το 2015 θα φτάσουν κάπου ανάμεσα στις 16 και τις 20.000. Την τελευταία εβδομάδα 1.240 αιτούντες άσυλο έφτασαν στη χώρα, οι περισσότεροι από την Συρία, όμως και αρκετοί από την Ερυθρέα και το Αφγανιστάν. Οι περισσότεροι από αυτούς πηγαίνουν στην Ορβηγία από άλλες χώρες του Σέγγεν, όμως τελευταία κάποιοι Σύριοι πρόσφυγες έφτασαν μέσω των συνόρων με την Ρωσία. Και στην ε, Νορβηγία υπάρχει μεγάλη πολιτική συνένεση για το ότι αυτή η κατάσταση θέλει μια κοινή ευρωπαϊκή λύση. Γι' αυτό παρακολουθούμε στενά τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για, την, ε, για το μηχανισμό έκτακτης ανάγκης και μετα, με, Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ε, ευθύνες μας και να εισέλθουμε στον πολιτικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργό μα, ε, Χόλμπεργκ, είχε συζητήσεις με την ε, καγκελάριο Μέρκελ πρόσφατα και οι πολλοί υπουργοί μας παρευρέθησαν σε ε, συνεδριάσεις, μεταξύ άλλων την εχθεσινή συνεδρία των Υπουργών Εσωτερικών. Πρόθεσή μας είναι να συμμετέχει και η χώρα μας εθελοντικά στον μηχανισμό μετακατάστασης και πανεκατάστασης. Πριν τις ε, θερινές διακοπές είχαμε συζητήσει το θέμα στο Κοινοβούλιο και ο αρχικό του Εργατικού Κόμματος πήρε την πρωτοβουλία για να οδηγηθούμε σε μια ευρύτερη συνένεση για το θέμα αυτό. Καταφέραμε λοιπόν να υπογράψουμε μια πολιτική συμφωνία για την συνεισφορά της Νορβηγίας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία και τις γειτονικές της χώρες. Υπήρχε γενική συνένεση για την ευθύνη που έχει και η Νορβηγία να συνεισφέρει στην ε, προσπάθεια αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, η Νορβηγία θα αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία και τις γειτονικές της χώρες κατά 27 εκατομμύρια ευρώ το 2015. Συνολικά, η στήριξη της ε, χώρας μας θα ανέρχεται στα 135 εκατομμύρια ευρώ φέτος και το 2016 θα προσθεθούν άλλα 27 εκατομμύρια ευρώ. Η Νορβηγία ενημέρωσε τον ε, υπατορμοστή των ΗΠΑ για τους πρόσφυγες ότι είναι έτοιμη να υποδεχτεί συνολικά 8.000 πρόσφυγες από τη Συρία από το 2015 μέχρι το 2017 και η ποσόστοση των ε, Σύρων προσφύγων που θα επαναγκατασταθούν θα αυξηθεί κατά 500 από δηλαδή 1.500 σε 2.000. Ε, οι δήμοι, οι κοινότητες και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις της ε, Νορβηγίας ε, κλήθηκαν να συνεισφέρουν στην άφηξη, την ενσωμάτωση και την εγκατάσταση των προσφύγων που φτάνουν στη χώρα. Ξέρουμε πως υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και ανάμεσα στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και στους πολίτες μας να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να ενταχθούν με επιτυχία οι Δήμοι οι οποίοι θα λάβουν περισσότερους πρόσφυγες από όσους τους ε, αναλογούν, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, θα λάβουν ε, περαιτέρω οικονομικές ενισχύσεις και επίσης θα υπάρχει επιπλέον ε, χρηματοδότηση για ενοικίαση στέγασης. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου η Νορβηγία με τη συνεισφορά δύο πλοίων στην Μεσόγειο διέσωσε πάνω από 7.000 πρόσφυγες και σκοπεύουμε να επεκτείνουμε αυτήν, να παρατείνουμε μάλλον αυτήν την ε, συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος επίσης των ε, εμπορικών ε, σκαφών στη διάσωση προσφύγων στη Μεσόγειο και τα νορβηγικά πλοία του εμπορικού ναυτικού έχουν συνεισφέρει σημαντικά. Η κυβέρνησή μας έχει στηρίξει ένα πρόγραμμα ασύλου στην Ελλάδα μέσω των ε, Norway Grants και μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επίσης, έχει γίνει πρόταση να ανακατανεμηθούν κονδύλια που θα αντιμετωπίσουν την ε, κρίση που διανύουμε. Επιπλέον, έχουμε εγκρίνει οικονομικές ενισχύσεις για την ε, πρώην Κυκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συνάντηση σήμερα και να σας εκφράσω την, το μεγάλο μου ενδιαφέρον για την συζήτηση που ακολουθεί. Ευχαριστώ κύριε Χένριξεν. Τελευταίος παρεμβαίνων της ημέρας, ο κ. Μάλια, της, οικονομικής, της ΕΟΚΕ, εισηγητής για γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Θέματα Μετανάστευσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας εκθέσω τις απόψεις της ΕΟΚΕ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΒΕ για την ευκαιρία αυτή και για το ότι δημιούργησε μια πλατφόρμα διαλόγου και συζήτησης. Πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογος, να συνεχιστούν οι συζητήσεις, διότι είναι σαφές πως πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μία νέα ε, αντιμετώπιση και να κινηθεί ενωμένη. Φυσικά έχει ασκηθεί έντονη κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να είμαστε σε θέση όχι μόνο να μείνουμε στα λόγια, να, να αναλάβουμε δράση. Πιστεύω πως αυτή η κρίση είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη και πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες είναι μια κρίση η οποία κινδυνεύει ε, να διχάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα γινόταν εάν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γινόταν εάν τα κράτη-μέλη ήταν μόνα τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ένα ψήφισμα την περασμένη εβδομάδα με ομοφωνία. Το ψήφισμα αυτό πιστεύω πως στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο μοιραζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δείχνει ότι πραγματικά είναι δυνατόν να υπάρχει ομόνια και ενότητα. Στο ψήφισμα αυτό ζητούμε αλληλεγγύη, ζητούμε αλληλεγγύη προς αυτούς τους μετανάστες οι οποίοι ε, αξίζουν προστασία, χρήζουν ασύλου και ζητούμε επίσης αλληλεγγύη με τα μεμονωμένα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα με τα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες πιέσεις σε αυτήν την κρίση καλούμε για μια γρήγορη ταχύτατη λύση στα κρατημέλη. Ε, φυσικά και στην Επιτροπή μας υπήρχαν διάφορες απόψεις και όμως ε, όλοι κατανόησαν ότι πλέον έχει έρθει η ώρα να δείξουμε στην πράξη τι σημαίνουν οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αρνητικές αντιδράσεις στην αντιμετωπίση της κρίσης. Είδαμε να κλείνουν σύνορα, να, ανεβαίνουν, να υψώνονται τείχη και καθυστερήσαμε πάρα πολύ να αντιδράσουμε θετικά. Βέβαια η χθεσινή συμφωνία ότι 160.000 ετούντες άσυλο θα επανεγκατασταθούν και θα διανεμηθούν σε όλη την επικράτεια της Ένωσης ήταν κάτι θετικό. Μην ξεχνάμε όμως το πόσο δύσκολο είναι ένα τέτοιο εγχείρημα. Βέβαια, αν δούμε χώρες όπως την Ιορδανία ε, ή την Τουρκία που έχουν να αντιμετωπίσουν εκατομμύρια προσφύγων, πραγματικά αξίζει να αναρωτηθούμε εάν αρκούν όλα αυτά που κάνουμε. Η ΕΟΚΕ έχει καταρτήσει αρκετές γνωμοδοτήσεις ε, σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα και με τους πρόσφυγες και εγώ ίδιος ήμουν πριν από δύο χρόνια εισηγητής για την ε, για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο μετανάστευσης στην Μεσόγειο. Μας πήρε πάρα πολλά χρόνια για να αποδεχτούμε και να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι πως αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού. Και στο παραπέντε έχουμε φτάσει να σκεφτόμαστε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Κατά την κατάρτιση της γνωμοδότησής μας, η οποία θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο, να σας πω, είχαμε διάφορες προκλήσεις ή τις συνήθεις ε, στην κατάρτιση μιας έκθεσης. Θα στείλουμε μια αντιπροσωπεία στη Σικελία, η οποία θα επισκεφτεί διάφορα κέντρα υποδοχής, θα μιλήσουμε με πρόσφυγες και θα συναντήσουμε ανθρώπους οι οποίοι ε, είναι στην πρώτη γραμμή της υποδοχής προσφύγων από την Frontex, συνοριοφύλακες και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. Για μας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, διότι χωρίς τη βοήθεια αυτών των τοπικών ε, ΜΚΟ και της κοινωνίας των ε, πολιτών δεν θα καταφέρναμε να είχαμε ως ε, κράτη-μέλη τη δυνατότητα, τις δυνατότητες που έχουμε τώρα. Θα ήμασταν πάρα πολύ περιορισμένοι. Φυσικά υπάρχουν και ευρωπαϊκά πλαίσια όπως η Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Γειτονία, η Συμφωνία για την Μεταγκατάσταση, όμως θα εστιάσουμε κυρίως σε δύο πτυχές. Στην κοινωνία των πολιτών, όπου θα δούμε πώς αυτή μπορεί να ενωθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική στην ε, πρώτη γραμμή της υποδοχής προσφύγων και η δεύτερη πτυχή πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών να ανταποκριθεί. Η κοινωνία των πολιτών βέβαια δεν έχει χρηματικούς πόρους και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνδράμει έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα αποτελεσματικά. Επίσης θα εστιάσουμε στην ένταξη. Κύρια προτεραιότητά μας βέβαια τώρα είναι να διαχειριστούμε αυτήν την κρίση με αποτελεσματικότητα. Αλλά βέβαια πρέπει να συζητήσουμε και το τι θα γίνει μετά, στο μέλλον, μετά την αποδοχή των ε, τον άσυλο. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να δεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσουμε άσυλο και μετά να τους αφήσουμε στην τύχη τους. Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως κινδυνεύσουν ξανά κινδυνεύσουν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευση και να είναι ευάλωτοι σε, σε διάφορα δεινά. Πρέπει να αποτρέψουμε μια δυσάρεστη κατάσταση και για τους ίδιους τους ετούντες άσυλο, να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να βρουν μια θέση στην κοινωνία η οποία τους δέχτηκε, να ενταχθούν σε αυτήν την κοινωνία και να μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτήν την κοινωνία. Είναι επομένως πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί κατάλληλη υποδομή γι' αυτό. Δυστυχώς οι εμπειρίες του παρελθόντος έχουν δείξει πως ε, δεν φτάνουν αυτά που κάνουμε, πως δημιουργούμε γκέτο και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ε, μετανάστες να συνεισφέρουν δημιουργικά στην κοινωνία μα, το οποίο θα βοηθήσει και τις ίδιες τις χώρες τις οποίες ε, εγκαθίστανται και οι πολίτες θα έχουν μια πιο θετική ακόμα εμπειρία με τους ε, πρόσφυγες. Όπως σας είπα, η γνωμοδότηση θα συζητηθεί το Δεκέμβριο και θα παρουσιαστεί τότε. Θα διεξαχθεί επίσης στις 15 Οκτωβρίου μία δημόσια κρόαση, όπου θα συζητηθούν συγκεκριμένα ζητήματα όπως η ένταξη στην αγορά εργασίας και τέλος το Δεκέμβριο θα γίνει η τελική συζήτηση και η ψηφοφορία της ε, γνωμοδότησης. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη τις δικές μας απόψεις και τη δική μας συνεισφορά για το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαριά. Έχουν περίπου δύο ώρες για συζήτηση, για ερωτήσεις, σχόλια. Να δώσω το λόγο στους εθνικούς βουλευτές και στους συναδέλφους στα μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κέσα από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Φοβούμε ότι πολλά από αυτά που άκουσα σήμερα διαπνεόταν από επιθυμία παραγωγής λύσεως. Δυστυχώς όμως πολλά από αυτά που υπόθηκαν δεν είναι ρεαλιστικά. Φοβούμαι ότι αυτό που συμβαίνει, κυρίως αναφορά την χθεσινή απόφαση, να υπάρχει υποχρεωτική με ειδική πλειοψηφία να επιβληθούν αποφάσεις που θα επηρεάσουν αρκετές χώρες που δεν θέλουν τέτοια απόφαση, ε, δημιουργείται κάτι σαν θάλαμο συμπίεσης σαν αποτέλεσμα και οι χώρες Στι χώρε αυτές θα αποφασίσουν τελικά οι ψηφοφόροι για τη λύση. Ανησυχώ τα μάλα λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο εκτελήσετε τα πράγματα. Και έχω ερώτηση. Υπάρχουν όρια, υπάρχει κάποιο όριο. Πώς, πόσοι μπορούν να έρθουν από καταπιεστικά καθεστώτα από τη Μέση Ανατολή ή την Αφρική. Μόνο εκείνοι που έχουν τα χρήματα να έρθουν. Αυτοί θα έχουν δικαίωμα να έρθουν ή μπορούν να έρθουν. Μήπως είναι οικονομική μετανά σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια κάποιος πρέπει να δείχνει κατανόηση ε, για τους πραγματικούς πρόσφυγες. Είναι πραγματικοί πρόσφυγες, αυτό είναι το ερώτημα. Και εξού και το επόμενο. Τι είναι πρόσφυγας, ποιος είναι ο ορισμός του πρόσφυγα σύμφωνα με τη σύμβαση του 1951 και σχετικά με τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειάζεται σαφέστερος ορισμός του πρόσφυγα. Τι είναι πρόσφυγας, ποιος είναι πρόσφυγας. Τελευταία ερώτηση. Οι τσιχαντιστές δεν αναφέρθηκαν καθόλου μέχρι τώρα. Θα είναι πολύ παράδοξη η κατάσταση αν ανακαλύψουμε ότι έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που θα μπορούσαν να καταφθάσουν και περνάει κρίσιμη φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση και διαλύεται όλο και περισσότερο, αποσυντίθεται και το έδειξαν οι ψηφοφόροι στο, στο ευρωβαρόμετρο ότι έχουμε έναν παράγοντα μείον 60 όσον αφορά την εμπιστοσύνη. Ερώτηση. Θα υπάρξει πραγματική ένταξη Μήπως θα έρθουν διάφοροι λαοί με διαφορετικούς νόμους, έθιμα και παραδόσεις που δεν θέλουν να ενταχθούν και να στερνιστούν τις ευρωπαϊκές αξίες που αναφέρονται εδώ επανειλημμένα, αλληλεγγύη κλπ. κλπ. Μήπως, ενδεχομένως λέω, δημιουργούμε ένα πρόβλημα που θα απορρίψουν οι ψηφοφόροι και θα τίνει να αποσυνθέσει την Ευρώπη αντί να την κάνει μια ισχύ, μια δύναμη πιο συνεκτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάσου. Ο κύριος Μπάτεν του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια απλή ερώτηση σε δύο τμήματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια εισαγωγή. Είπε ο Κιβές, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών του, της Βουλής των Κοινοτήτων είπε δύο πράγματα. Αναφέρθηκε στους μετανάστες και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα σχέδιο που μπορεί να πουλήσει στο εκλογικό σώμα. Χαίρομαι που ανέφερε του μετανάστε, γιατί στην Επιτροπή αναφέρθηκαν πολλά για πρόσφυγε και τούντε άσυλο. Και η Σύμβαση των 51 αναφέρει επακριβώ τα κριτήρια για το ποιο είναι πρόσφυγα. Και πολλοί ή τεράστια πλειοψηφία εκείνων που είναι στι πύλε τη Ευρώπη δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Δεν είναι πρόσφυγε, είναι μετανάστε και παράνομοι μετανάστες. Μετά είπε, υποθέτω ότι εννοεί την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα σχέδιο που να μπορεί να πωλήσει στο εκλογικό σώμα. Οι πολιτικοί πάντα θεωρούν ότι αν μπορώ να εξογήσω μη δημοφιλείς πολιτικές ε, δεν μπορώ να τις πουλήσω στην, στο λαό. Δεν μπορεί να πουλήσεις κάτι στο λαό αν δεν το θέλει και αν τα καταφέρεις, δεν είσαι πολιτής αλλά κάποιος κομπιναδόρος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλουν ατέρμονα κύματα μετανάστευσης μαζικής. Είδαμε διαδηλώσει όλη την Ευρώπη επίσης. Στο πολιτικός ορθό BBC δεν το δείχνω αυτό. Είναι ηρωνικό ότι πρέπει να πας στο RT που είναι το ρωσικό κανάλι προπαγάνδας για να μάθεις την αλήθεια. Και δείξαν εκεί τις διαδηλώσεις στην Ευρώπη χθε στην Επιτροπή εδώ η Ουγγαρία επεκρίθη διότι η Ουγγρική κυβέρνηση είχε το θάρρος να ρωτήσει τους πολίτες τι θέλουν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να το κάνει αυτό είναι, διότι ξέρει καλύτερα από τους πολίτες τι θέλουν. Και κάποιοι από τους ελάχιστους που μίλησαν λογικά στην κρίση ήταν ο Βίκτορ Ορμπάν και χαίρομαι που είδα ότι ο Ούγγρος ε, Επίτροπος στήριξε τη χώρα του. Αυξάνονται οι μετανάστες και έχουν συγκεκριμένη νοοτροπία. Και βλέπουμε ότι δεν είναι μετανάστευση αυτό που γίνεται, είναι ε, εισβολή. Κοιτάξτε τη στάση των νέων στο Καλέ και την Ουγγαρία. Δεν ζητάνε ευγενικά να τους επιτραπεί είσοδος, διότι διώκονται στις χώρες τους, απαιτούν είσοδο. Είναι επιθετικοί, είναι υπερφύαλοι. Όσο τους αφήνουμε αυτούς να μπαίνουν, όλο περισσότεροι θα καταφθάνουν. Ο κ. Μάλια είπε ότι πού θα ήταν το πρόβλημα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχε. Πιθανότατα αυτό το πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Διότι η κυρία Μέρκελ, όπως είπαμε, κάλεσε όσους ήθελαν να έρθουν να έρθουν στη Γερμανία. Και τώρα δρέπει τους καρπούς της πράξης. Και λόγω των ανοιχτών συνόρων του Σέγγεν αυτοί ξέρουν όταν πατήσουν σε μια χώρα μπορούν να μπουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη και να φτάσουν μέχρι το καλέ. Και βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες. Αυτό αναφέρθηκε ήδη. Θα ήταν πολύ λογικότερο αν ζητούσαν άσυλο σε μουσουλμανικές χώρες και ακολουθούσαν άλλη κατεύθυνση. Δύο απλές ερωτήσεις έχω τώρα προς την Επιτροπή. Δέχεται η Επιτροπή ότι η τεράστια πλειοψηφία αυτών που προσπαθούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πρόσφυγες και άσυλο, αλλά μετανάστες και παράνομοι μετανάστες. Και γι' αυτό η πολιτική μας θα πρέπει δόντως να το αντικατοπτρίζει αυτό. Δεύτερον, δέχεται η Επιτροπή ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάθε διπλωματική πίεση και πρακτικά μέσα συντονισμένα μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις Ευρώπης, ούτως ώστε να ασκηθούν πιέσεις επί των πλουσιωτάτων μουσουλμανικών χωρών του κόλπου, Φερρυπίν, που θα μπορούσαν να τους δεχτούν αυτού και να τους φιλοξενήσουν. Είναι σε πολύ καλή τη θέση να το κάνουν. Θα ταιριάζαν καλύτερα, θα εντασσόταν καλύτερα, θα ήταν καλύτερο και για αυτούς και για μας. Και μπορούν να το στηρίξουν οικονομικά γιατί είναι πάμπλουτες. Ευχαριστώ κύριε Μπάτεν. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάποιος που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, οπότε η ερώτησή σας αφορούσε το πρωινό, την πρωινή συνεδρίαση τώρα. Ο κύριος Κόλσο. Από τη Λετωνία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα συνεχίσω τα λετωνικά, Λίγο μιλητής. Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλούμε και πάλι για τις συνέπειες. Τι θα κάνουμε με την κοινωνική ένταξη, τι άλλα μέτρα θα αναλάβουμε κτλ. Αλλά σε εθνικό και τοπικό επίπεδο πρέπει ακόμα να μιλούμε για τις αιτίες της κρίσεως, που είναι το οργανωμένο έγκλημα το οποίο αυτή τη στιγμή το εξετάζουμε στο μεσογειακό του πλαίσιο αλλά πηγαίνει πολύ πέραν αυτού είναι εξαιρετικά δραστήριο και εντός των ευρωπαϊκών σύνορων είδαμε τι έγινε και στα αυστρο σύνορα το οποίο σημαίνει αυτομάτως την συμμετοχή Ευρωπαίων πολιτών στα οργανωμένα αυτά εγκληματικά δίκτυα. Και επομένω θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικαιροποιήσει τους ποινικού της κώδικες και να αυξήσει τις ποινές για τα δικήματα που έχουν σχέση με τη διακίνηση ανθρώπων. Σε εθνικό επίπεδο θα είναι δύσκολο να καταπολεμήσουμε τα εγκληματικά αυτά δίκτυα, διότι είναι διασυνοριακά και θα πρέπει να ενέχεται και η Ευρωπόλ στην προσπάθεια αυτή. Αλλά σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ανοιχνεύσουμε τους υπεύθυνους που στην τελική ανάλυση είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε τα αίτια της μετανάστευσης, λέει ο μιλητής. Και όταν ακούω ότι η Europol δεν έχει επαρκείς πόρους για να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα, ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα κατασχεθέντα ποσά για να ενισχύσουμε την Europol και τους άλλους φορείς. Γι' αυτό ζητώ την ε, κατεπίγουσα επικαιροποίηση των ποινικών κωδίκων των κρατών μελών και των εθνικών διατάξεων. Σας ευχαριστώ κυρία Wimberg. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σας πω δύο λόγια για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, στη Σουηδία. Έχουμε περί τους 7.000 που προσέρχονται κάθε εβδομάδα. Διερωτάται κανείς αν υπάρχει τέλος. Και συζητούμε εδώ για το δουμπλίνο στη Σουηδία ε, αυτή τη στιγμή ε, χρειάζεται τόσος πολύς χρόνος για να ζητήσει κανείς άσυλο που τους παρέχουμε δωρεάν εισιτήριο τρένου στη Βόρεια Σουηδία και μετά περνούν στη Φιλανδία διότι απλούστατα η διοικητική διαδικασία είναι εξαιρετικά μακροσκελής. Η ένταξη έχει αποτύχει και αποτυγχάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν φαντάζομαι ότι πρόκειται να βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον. Επίσης, παρατηρούμε μια ασάφεια σχετικά με την ανάλυση των αιτιών του φαινομένου. Ακούμε και ακούσαμε και πρόσφατα ότι δεν λαμβάνουμε βοήθεια χρηματική ε, για τα κέντρα υποδοχής. Εάν όμως οι άνθρωποι είναι τόσο απελπισμένοι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε να βοηθήσουμε τους περισσότερους ανθρώπους που μπορούμε στις περιοχές που μπορούμε αντί να ψάξουμε να ε, ε, ρυθμίσουμε ή να βοηθήσουμε τις τύχες τους ε, απέναντι από τη Μεσόγειο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προσδοκίες βοήθειας για τους ανθρώπους αυτούς. Ακούσαμε από το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα ότι έχουν γίνει αιτήματα επίγουσας βοήθειας, ότι θέλουν να μοιράσουν ε, κουπόνια σύντησης. Ε, πρέπει να δούμε τα αίτια του πράγματος αυτού. Γνωρίζουμε πόσα εκατομμύρια ανθρώπων περιμένουν στην Τουρκία για να περάσουν απέναντι. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό με κάποιες κλίδες κατανομής. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στα βαθύτερα αίτια. Ευχαριστούμε την κυρία Βίνμπεργκ. Ο κύριος Ζαμίτε Ντίμε της Μάλτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα να είμαστε εδώ. Όταν διοργανώθηκε αυτή η συνάντηση δεν είχαμε φανταστεί βέβαια ότι θα υπήρξε παράλληλη έκτακτη σύνοδος σχετικά με το θέμα αυτό, το πολύ σημαντικό και σοβαρό αυτό θέμα της μετανάστευσης. Και όλοι εδώ εξετάζουμε το θέμα υπο, ο καθένας υπό την ε, εθνική του οπτική γωνία. Εγώ να σας προσφέρω τη δική μας. Από το 2002 καταγράφουμε μεταναστευτικές εισρωές από τη Βόρεια Αφρική και ιδιαίτερως από τη Λιβύη. Στην πραγματικότητα οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική, από τη Σομαλία, από την Ερυθρέα. Και, για πάρα πολλά χρόνια είχαμε 2.000 και πλέον προσελεύσεις κάθε χρόνο. Αυτό πρέπει να το δει κανείς βεβαίως στα πλαίσια του μεγέθους της χώρας. Μιλούμε για μια χώρα με 420.000 κατοίκους και μια πυκνότητα πληθυσμού άνω των χιλίων ανθρώπων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. χιλίων τρακοσίων. Εμείς τονίζουμε συνεχώς και υπογραμμίζουμε συνεχώς ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Γιατί δυστυχώς για μια χώρα σαν τη δική μας, αλλά και για την Ιταλία και για την Ελλάδα, Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που επισημαίνουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα, αλλά δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, διότι άλλες χώρες δεν έχουν κάνει τίποτε στην πραγματικότητα, λέγοντας, αναλαμβάνοντας την απλή τοποθέτηση, ότι κοιτάξτε, δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Και κάποια τραγικά συμβάντα των τελευταίων μηνών, η απώλεια της ζωής 2.500 και άνω ανθρώπων στην προσπάθειά του να προσέλθουν στην Ευρώπη. Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν, οι τραγικές αυτές εικόνες, έχουν αυξήσει αυτήν την αίσθηση του κατεπήγοντος. Και αυτό είναι που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε με αποτελεσματικότητα και ενδελεχώς τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας και θα πρέπει να δούμε εξεταστικά, ε, προσεκτικά με τη διάκριση μεταξύ ενός πρόσφυγα που διαφεύγει από μια κατάσταση πολεμική συγκρούσεως στη χώρα του και ενός οικονομικού μετανάστη. Έχουμε ένα μέσο ποσοστό άνω του 20% στη διαχείριση φακέλων ετούντων άσυλο, δηλαδή το ψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχόμαστε ότι στη σημερινή σύνοδο η επανεγκατάσταση των 160 αυτών χιλιάδων θα είναι ένα μικρό βήμα αλλά βασικά ευχόμαστε ότι όλα τα μέσα στα οποία θα υπάρξει συμφωνία θα υλοποιηθούν, θα τεθούν σε εφαρμογή από την επόμενη αμέσως ημέρα της συμφωνίας αυτής. Γιατί αυτό είναι μια δοκιμή αξιοπιστίας αυτή τη στιγμή για τις αρχές που υποστηρίζουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Άννα Γκόμες, ε, της Επιτροπής Λίμπε. Θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά ότι είμαι μία από τις ευρωβουλευτές εδώ που ζητά να επιβληθούν κυρώσεις στην Ουγγαρία για τη συμπεριφορά της. Διότι πιστεύω πως η στάση της Ουγγαρίας αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση δεν πρεσβεύει τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν δεν με απατάει μνήμη μου, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Σύμβαση για τους πρόσφυγες είχε γίνει για Ευρωπαίους. Εκείνοι ήταν οι πρόσφυγες, εμείς ήμασταν οι πρόσφυγες. Και συμφωνώ με την συνάδελφο από την Νορβηγία που επέστησε την προσοχή μας στο ότι αυτή είναι μια νέα εποχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη. Και από την άλλη, όπως είπε και ο συνάδελφος από τη Μάλτα, είναι κάτι που δεν είναι καινούριο, γίνεται εδώ και καιρό. Και πρόσφυγες και μετανάστες έρχονται στην Ευρώπη. Είμαστε μία ήπειρος που αποτελείται από πρόσφυγες και μετανάστες. Ο κόσμος έχει δημιουργηθεί από μεταναστευτικές ε, ροές, από κόσμο που φεύγει από ένα μέρος και πάει στο άλλο. Δεν άρχισε το 2002 το πρόβλημα. Υπάρχουν ευθύνες και η άρνηση ορισμένων χωρών να τις αναλάβουν αυτές τις ευθύνες έχει κάνει τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν προερχόμαστε από μία ήπειρο η οποία έχει γεννήσει μετανάστες. Εγώ είμαι από την Πορτογαλία και η Πορτογαλία λόγω της πολιτικής λιτότητας που έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δημιουργήσει 485.000 μετανάστες. Μας έχουν φύγει λοιπόν περίπου μισό εκατομμύριο ε, άτομα, τα οποία χρειαζόμασταν γιατί είναι καταρτισμένα άτομα, είναι μορφωμένα, όπως και οι Σύριοι οι οποίοι έρχονται εδώ στην Ευρώπη, οι οποίοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους, όχι επειδή ε, το θέλουν, αλλά επειδή αναγκάστηκαν, αναγκάστηκαν από τη βιαιότητα που επικρατεί και στη Συρία και στο Ιράκ. Και το λέω αυτό γιατί πριν από δέκα μέρες ήμουν εκεί, ήμουν στα σύνορα της Συρίας με το Ιράκ και μπορώ να σας πω ότι οι κυβερνήσεις μας έχουν αποτύχει και προς ε, εκείνους τους ανθρώπους και προς τα εμάς. Δεν έκαναν τίποτα για να κατοπολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος και δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικοί για την επίλυση των ε, σειράξεων, όπως θα έπρεπε να είναι. Ήμουν εισηγήτρια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για το θέμα αυτό και πρέπει να σας πω στο θέμα της Λιβύης ότι δεν, μία μόνο κυβέρνηση έμεινε μετά από όλα τα γεγονότα η οποία κυβέρνηση που έμεινε όρθια δεν έκανε τίποτα από αυτά που έπρεπε να κάνει. Ούτε μεταρρυθμίσεις έκανε, ούτε διαρθρωτικές, ούτε σε άλλους τομείς, ούτε κατάφερε να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές. Τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε. Εάν δεν υπήρχε τάξη στην ε, Λιβύη δεν θα υπήρχαν και αυτά που βλέπουμε, τα οποία βλέπουμε τώρα. Και στην ουσία αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι άνευ προηγουμένου. Σπαταλάμε πόρους για ανούσια πράγματα, πόρους οι οποίοι εξαφανίζονται εκεί, ενώ θα έπρεπε να κάνουμε τελείως ε, διαφορετικά πράγματα. Θα έπρεπε να καλωσορίζουμε πολύ περισσότερους πρόσφυγες στην Ευρώπη και να είμαστε πολύ ε, πιο αποτελεσματικοί στο τι γίνεται εκεί, από εκεί που ξεκινάνε. Και αναφέρομαι στο, στην ε, καταπολέμηση των ε, αιτιών, Κατα, αναφέρομαι στην, στο Ισλαμικό κράτος, στους ε, τζιχαντιστές. Και να απαντήσω τώρα και σε αυτούς που ανέφεραν τον τζιχαντισμό. Ξέρετε ποιοι είναι τζιχαντιστές στην Ευρώπη, οι δικοί μας, οι Ευρωπαίοι. Δεν χρειάζεται ο τζιχαντιστής να κάνει αυτό το απέσιο ταξίδι στην Ευρώπη. Όχι, ταξιδεύουν με πλαστά έγγραφα. Και αυτό δείχνει πως έχουμε αποτύχει παντελώς στο έργο μας. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες και για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει θεμελιωδώς η πολιτική μας. Διότι εάν δεν προστατεύσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη τώρα, δεν θα μπορέσουμε μετά να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Και μην ξεχνάτε ότι εκτός από τους πρόσφυγες έχουμε ανάγκη και από μετανάστες. Ο κύριος Λέγκενι από την Ουγγαρία έχει τώρα το λόγο, αν προφέρω καλά το όνομα του λέει η πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μένει πολύ χρόνος από ό,τι βλέπω και ήθελα να αναφέρω τρία στοιχεία. Το κόμμα των σοσιαλιστών ε, της Ουγγαρίας θεωρεί ότι το Δουβλίνο έχει αποτύχει. Δεν είναι ένα επαρκές πλαίσιο για να αντιμετωπίσει τη σημερινή κατάσταση. το πλαίσιό του θα μπορούσε να φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ κατώτερο των ροών που έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο σύστημα πρώτον. Δεύτερον, θεωρούμε ότι αυτή η μάζα των ανθρώπων έχουν φύγει από τις χώρες τους, από όπου και να προέρχονται, από τη Συρία, το Λίβανο, την Ιορδανία, μπορούμε να προσθέσουμε εκείνους που έρχονται από το Αφγανιστάν. Λόγω της ε, δυσμενούς κατάστασης που επικρατεί στις χώρες τους. αν θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των κέντρων υποδοχής σε εκείνες τις χώρες από τις οποίες περνούν, θα μπορούσαμε να μειώσουμε λίγο την εισρωή για την Ευρώπη. Τώρα για τα θέματα παγκόσμιας γεωπολιτικής μπορούμε να πούμε πολλά, για ορικά καύσιμα, για άλλα πράγματα, αλλά ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος και κημητήριος μοχλός είναι η ISIS. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την καταπολεμήσουμε για να εξομαλύνουμε την κατάσταση στη Συρία. Ε, σας ευχαριστώ. Η κυρία Άτκινσον από την Επιτροπή Λίμπε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπατριώτες μου που ήρθαν εδώ. Όπως βλέπετε κύριοι, ήρθατε στο άντρο των θηρίων. Τίποτα δεν θα γίνει σύντομα και χαιρετίζω τον εκπρόσωπο του Βίκτορ Όρμπαν, τη κυβερνήσεω του Βίκτορ Όρμπαν από την Ουγγαρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τεράστια πλειοψηφία του λαού υποστηρίζει αυτά που κάνατε. Και πολύ συχνά χρησιμοποιείτε μία φράση εδώ. Αλληλεγγύη. Δείχνετε αλληλεγγύη. Σέβεστε τις αξίε των συνθήκων που υπέγραψαν οι λαοί, ψώνοντα τους φράχτες. Έχω ερώτηση. Απευθυνόμενη προς τον κ. Φανσουάντι Κώστα. Ήμουν η μόνη πολιτικός του Ηνωμένου Βασίλειου που συναντήσε το Δήμαρχο του Καλέ πέρσι και συμφωνήσαμε επί πολλών. Θα επαναλάβω την ερώτηση που έθεσα το πρωί, διότι δεν απαντήθηκε. Σύμφωνα τη Σύμβαση του Δουβλίνου, μπορούμε να κρατήσουμε και να απελάσουμε εκείνους που είναι εγκληματίες και όχι μετανάστες, είναι εγκληματίες. Γκρεμίζουν τους φράχτες, ε, μπαίνουν στο τούνελ και επηρεάζουν την οικονομία της κομιτείας του Κέντ και είναι εγκληματίε διότι εισβάλλουν στα φορτηγά. Γιατί τους συλλαμβάνετε, γιατί δεν κρατούνται, γιατί δεν απελάβνονται. Είναι η ερώτησή μου. Uh, η κυρία Καρίνα Όλσον. Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε, εμάς από το Εθνικό Κοινοβούλιο, να παραστούμε στη σημαντική αυτή συνάντηση. Είμαι σοσιαλδημοκράτης από την Σουηδία και είναι τιμή για μένα, αλλά είναι σημαντική ε, επίσης τιμή να είμαι στην αίθουσα Αναλίντ που πάντα υποστήριζε τα ανθρωπίνα δικαιώματα και θα έπρεπε να είναι η αφετηρία των σημερινών συζητήσεων αυτό. Και αυτό δεν βγαίνει από τη συζήτηση τόσο ξεκάθαρα είναι πολύ οξία η συζήτηση. Η κατάσταση είναι προβληματική, πρέπει να σώσουμε ζωές. Χρειάζεται προετοιμασία. Ταυτόχρονα πρέπει να συζητήσουμε εξωτερική πολιτική. Ειρηνευτικά μέτρα. Πολιτική αναπτυξιακή. Να και στηρίζουμε και την ύπατη αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σουηδία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν και το δικαίωμα ασύλου ξεφεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από το πόλεμο, παιδιά ξεφεύγουν μεταξύ αυτών και προβλέπουμε στη Σουηδία ότι πάνω από 80.000 ετούντες άσυλο θα καταφτάσουν φέτος. 20.000 από αυτούς θα είναι παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους. Και έχουμε μακρά παράδοση υποδοχής παιδιών που ταξιδεύουν μόνα τους στη Σουηδία. Έχουμε δεχτεί σημαντικό αριθμό από τη Φιλανδία πριν από πολλά χρόνια. Έχουμε μακρά παράδοση να βοηθείας προς εκείνους που ξεφεύγουν τον πόλεμο και ιδιαίτερα προς τα παιδιά. Είναι μια κοινή ευθύνη αυτή. Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη και αυτό που έχουμε είναι μια καλή αρχή. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη για την οποία θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι Προφανώς υπάρχουν πολλά μέτρα που απαιτούνται ανάλογα με την αντιμετωπιζόμενη κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεφεύγουν από τον πόλεμο τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα δημιουργήσουμε νομικές διόδους μετανάστευσης. Όπως είπε κάποιος χρειάζεται και αναθεώρηση η σύμβαση του Δουβλίνου. Θα πρέπει να αυξηθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών. Όταν μιλάμε για εθνική διάσταση και τοπική διάσταση και περιφερειακή διάσταση Όλα αυτά αποτελούν τμήμα των συζητήσεων που γίνονται στις χώρες μας. Δεν μιλάμε για αλληλεγγύη μεταξύ χωρών μόνο, αλλά και αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων επιπέδων σε μια χώρα. Όλοι θα αναγνωρίσουμε ότι ξεκινάμε πάντα τη συζήτηση από μετανάστευση και καταλήγουμε σε ολοκλήρωση. Για τα παιδιά, πρόσβαση στην υγεία, στη μέρημνα, ε, στη δυνατότητα να πάνε σχολείο, κάπου να μπορούν να ζήσουν. Ε, δηλαδή και όλα αυτά αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών και την προστασία των δικαιωμάτων παιδιών. Οι ενήλικες βέβαια θα πρέπει να προσπαθούν, να μπορούν μάλλον να, να ζήσουν. Πρέπει να δούμε ποια καλά παραδείγματα υπάρχουν που έχουν πετύχει συστήματα πάνω σε αυτό. Όσον αφορά το δικαίωμα ασύλου, χρειάζεται πράγματι χρόνο στη Σουηδία για τη χορήγηση ασύλου. Πρέπει να επιταχύνουμε τι διαδικασίε. Όμω εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, την αξιολογούμε, κάνουμε σωστή αξιολόγηση εξετάζουμε τις λεπτομέρειες κάθε αιτήματο ε, ασύλου. Δεν είναι ότι αφήνουμε οποιανδήποτε να μπει, όχι, εξετάζουμε προσεκτικά τις αιτήσει ασύλου, ε, έτσι χειριζόμαστε το θέμα. Σαφώς υπάρχει μια κοινή ευθύνη όλων μας και αν εξετάσουμε την κατάσταση θα βρούμε και καλά και κακά παραδείγματα. Έχουν 500 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεχόμαστε ένα εκατομμύριο. Είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Αν δείτε τι γίνεται στην Τουρκία, υπάρχουν περισσότεροι πρόσφυγες σε αυτή τη χώρα από ό,τι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη τις αναλογίες όταν συζητούμε το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Όλσον. Ο κύριος Τεσελής από την Ουγγαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, κάποιες πτυχές και ελπίζω ότι θα κατανοήσετε τα ουσιαστικά στοιχεία του μηνύματος που θέλω να σας στείλω. Ίσως δεν γνωρίζετε το πρόσφατο παρελθόν της Ουγγαρίας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η Ουγγαρία δέχτηκε τους πρόσφυγες από την Ελλάδα που ξέφευγαν από τον εμφύλιο στην Ελλάδα. Το χωριό του Μπελογιάννης δέχτηκε 400 οικογένειες στην ε, Ουγγαρία. Ανήκει στην εκλογική μου περιφέρεια και ο, το, ο νέος νόμος της Ουγγαρίας επέτρεψε στην ε, κοινότητα την ελληνική να έχει και εκπρόσωπο στην Εθνοσυνέλευση. Δεν θα το γνωρίζετε ίσως, δεν θα γνωρίζετε τι συνέβη κατά τη διάρκεια του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Δέχτηκε εκεί η Ουγγαρία όλους τους πρόσφυγες που προερχόταν από την πρώην Γιουγκοσλαβία ανεξάρτητα της εθνότητάς τους ή της θρησκείας τους. Το πρώτο κέντρο υποδοχής στη Νέα Δημοκρατία μετά το 1990 κατασκευάστηκε στο Μπίτσκε στην Ουγγαρία Εκεί ήμουν δήμαρχος εγώ για δύο θητείες. Εκπροσωπώ την κοινότητα σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, ε, ε, μάλιστα βοηθήσαμε χιλιάδες πρόσφυγες. Πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω, όλα άλλαξαν έκτοτε. Αυτοί που φτάνουν στην ε, Ουγγαρία δεν δέχονται πια τη βοήθειά μας. Είναι ε, βίαιοι, υπερφύαλοι, ε, αλαζονικοί. Ε, ε, και ε, φέρονται άσχημα στους ντόπιου. παραβιάζουν πόρτες και το έκαναν αυτές τις τελευταίες ημέρες. Πριν βοηθούσαμε κόσμο που αντιμετώπιζε πραγματικό κίνδυνο. Σήμερα το 7% των ετούντων άσυλο είναι αυτοί που ξεφεύγουν από πραγματικό κίνδυνο. Σκεφτείτε το αυτό. Μήπως πρόκειται περί μεταναστών που ε, ε σας παραπλανούν από τον πραγματικό κίνδυνο. Αποσπούν την προσοχή σας. Υπάρχει πραγματικά σύγκρουση στην Ουκρανία και αυτή είναι μια κατάσταση που μας ανησυχεί πολύ. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία σέβεται τον νόμο και αυτή απειλείται από αυτό το φαινόμενο. Μη, θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί κανόνες. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι η Ουγγαρία δεν έκλεισε τα σύνορά της. Έκλεισε τα σύνορά της τα πράσινα, τα ανοιχτά της σύνορα, συγγνώμη μάλλον. Ενισχύουμε την προστασία, την νομική προστασία τη φυσική προστασία παρέχουμε που απαιτείται ε, μέσω ισχυροποίησης των ανθρωπίνων πόρων. 200.000 άνθρωποι πέρασαν παράνομα τα σύνορα της Ουγγαρίας και 175.000 ετούντες άσυλο καταχωρήθηκαν. Τούτου λεχθέντος η Ουγγαρία δεν είναι μια χώρα της πρώτης γραμμής, front line, δεν αποτελούν αντικείμενο νέας πρωτοβουλίας. Γιατί? Ο κύριος Ασνάρ του Ισπανικού Κοινοβουλίου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την προηγούμενη παρέμβαση του συναδέλφου από το Εθνικό μας Κοινοβουλίο. Εμείς υποφέρουμε, επιτρέψτε μου τον όρο, πολλά χρόνια τώρα, προσπαθώντας να ανταποκριθούμε αλληλέγγυα στο πρόβλημα. Αλλά επιτρέψτε μου μία παρατήρηση σχετικά με αυτά που συζητούμε από το πρωί. Σχετικά με το πολύ σοβαρό πρόβλημα, ίσως την πιο μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Προσπαθεί η Ευρώπη να ανταποκριθεί. Ίσως με το, όχι με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ίσως όχι με τον πιο ευλαβικό τρόπο αν θέλετε να το πω έτσι. Αλλά η Ευρώπη, τα θεσμικά μας όργανα, οι φορείς προσπαθούν, προσπαθούν όπως μπορούν να ανταποκριθούν με αλληλεγγύη. Και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα το καταφέρουν. Ακούσαμε όμως για την κυρία Γκόμες που μίλησε για δύο πτυχές. Εκείνους τους ετούντες άσυλο που φτάνουν στο έδαφος μας και την άλλη πτυχή που δεν είναι λιγότερο σημαντική. Τι συμβαίνει μέχρι να φτάσουν. Όλο αυτό το μαρτύριο που πρέπει να περάσουν μέχρι να φτάσουν εδώ. Οι φυστάμενοι επιθέσεις, και εκμετάλλευση κάθε είδους που δεν μπορούμε ούτε καν να τη φανταστούμε. Εμείς πράγματι έχουμε αυτή την υποχρέωση, την ανθρωπιστική και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε όσο πιο αλληλέγγυα μπορούμε. Όμως θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μόνη της εδώ. Δεν, όμως, δεν μιλούμε για τα 160.000 που ζητούν προστασία μιλούμε για πολλές ακόμα εκατοντάδες χιλιάδων που τις ερχόμενους μήνες και χρόνια θα χτυπήσουν την πόρτα μας. Και έχω την εντύπωση ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση η Ευρώπη είναι πολύ μόνη της. Και ρωτώ, αυτό το πρόβλημα είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν κάτι εδώ να πούν. Η Αραβική Λίγκα δεν έχει κάτι εδώ να πει όπως είπε και ο συνάδελφος που μίλησε νωρίτερα, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί. Και το δεύτερο που θέλω να σημειωθεί είναι το εξής. Καλείται η Ευρώπη να ηγηθεί και σε παγκόσμια κλίματα ακόμα σε εξωτερικά θέματα. Και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση εδώ, και να ασκήσουμε αυτόν τον ηγετικό ρόλο θα έπρεπε στο μέτρο του δυνατού μέσω διαπραγμάτευσης να συνεργαστούμε με άλλες υπερεθνικές οργανώσεις που αναφέρουμε αλλά και άλλες όχι κοντινές στα σύνορά μας αναγκαστικά αλλά κοντινές εδαφικά στις χώρες προελεύσεως αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που θέλουν να φύγουν από εκεί. Αυτήν την, αυτόν τον ηγετικό ρόλο πρέπει, πρέπει να τον αναλάβουμε και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Τώρα, είναι σίγουρο ότι με κάποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε με αυτές τις ελλειπείς προσπάθειες που κάνουμε. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική ως Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι ναι δικό μας το πρόβλημα, αλλά είναι και παγκόσμιο πρόβλημα και πρέπει να συμμετάσχουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε τον κύριο Αφινάρη. Ο κύριος Βάσκεθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλό απόγευμα σε όλους. Θα είμαι πολύ σύντομος διότι ε, συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφο μόλις μίλησε και θα αναφερθώ στο άλλο, στην άλλη πτυχή. Ότι δηλαδή δεν έχουμε ούτε αρκετή Ευρώπη στην Ένωση, ούτε αρκετή Ένωση στην Ευρώπη. Το είπε στις 9 του μηνός ο πρόεδρος Γιούγκερ, ότι η κρίση των προσφύγων πρέπει να είναι εφαλτήριο και για λόγους ανθρώπινης αξιοπρέπειας το δικαίωμα στο άσυλο δεν μπορεί παρά να είναι πρώτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπαν όλοι. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Και αυτό το τονίσαμε στις συζητήσεις ολόκληρη την ημέρα. Προφανώς με κάποιες αποχρώσεις. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ στα πλαίσια της μεταναστευτικής κρίσης. Δηλαδή ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στο οποίο αναφερθήκαμε στις συζητήσεις της πρωινής και επί του οποίου το Συμβούλιο είχε κάποιες συστάσεις για τους έλεγχους των εξωτερικών συνόρων που πρέπει να υποβληθούν πριν το τέλος του έτους. Δεν ξέρω αν κάποιος θα μπορούσε να απευθυνθεί στους αρμόδιους, στο κύριο Ντεκώστερ, δεν ξέρω κάποιο άλλο μέλος να διαβιβάσει την ερώτηση προς την Κομισιόν, δηλαδή ποια μέτρα σκοπεύουν να συμπεριλάβουν στην υφιστάμενη δέσμη των εφιών αυτών μέτρων στην αναθεώρηση που σκοπεύει, σκοπεύει να υποβάλει για να εφαρμοστεί το έτος 16. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάσκε. Στον κύριο Ντεκώστα θα δώσω το λόγο στο τέλος της συζητήσεως. Μπορείτε να στείλετε και γραπτό τις ερωτήσεις σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εκπροσωπεί την Επιτροπή των Περιφερειών και στο Ντεκώσταρ. Συνάδελφος της Επιτροπής Λίμπε, η κυρία Αναλυστίνη έχει το λόγο. Ε, thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υποθέτω ότι το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη αυτή την πρόκληση είναι βασικό ερώτημα. Αυτή τη στιγμή η πίεση είναι στις χώρες. Όμως η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη ενοποίηση έτσι ώστε να μπορέσει πιο αποφασιστικά και πιο ενεργά να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Η Άννα Γκόμες το περιέγραψε πολύ καλά. Και το επόμενο βήμα, η επόμενη πρόκληση είναι η πρόκληση της ένταξης, διότι εκείνοι που είναι ήδη εδώ χρειάζονται μία ολοκληρωμένη ολιστική προσέγγιση για την ε, ένταξη. Όπως πολύ σωστά υπόθηκε, ζούμε σε μία νέα εποχή και αυτά τα θέματα μπορούμε να τα λύσουμε μόνο εάν δράσουμε μαζί ως Ένωση και εάν ε, είμαστε πιο δραστήριοι και οι πολιτικές μας είναι πιο ολιστικές. Επίσης αυτό είναι κάτι που αναμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι μόνο. Ακούμε περισσότερη κριτική, αλλά λιγότερες προτάσεις και αυτό είναι που χρειαζόμαστε, οι προτάσεις. Το πρωί ακούσαμε τις απόψεις της Frontex, αλλά αυτά είναι μόνο τα μέτρα του πρώτου σταδίου. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε σε βάθος χρόνου, δεκαετιών, στην Εστονία, την πατρίδα μου. Έχουμε 400.000 μετανάστες από τη Ρωσία και είμαστε μια χώρα λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκων. Καταφέραμε να τους εντάξουμε τους μισούς από αυτούς και γλωσσικά και ε, να τους κάνουμε εστονούς υπηκόους, αλλά τους άλλους μισούς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τους εντάξουμε. Δεν έχουν ενταχθεί. Γι' αυτό λοιπόν αυτό σκεφτείτε το σε ευρωπαϊκή διάσταση. Η δική μου γενιά είναι γενιά παιδιών πολέμου και 60 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υπήρξαν πρόσφυγες. Η δική μου χώρα για παράδειγμα χρωστά ευγνωμοσύνη στη Σουηδία η οποία δέχτηκε δικούς μας πολίτες ε, το 1944 και αυτό είναι ένα επιχείρημα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και σήμερα σε συζητήσεις και σε αυτούς που είναι διχασμένοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι αξία ιστορική και είναι κάτι που μας βοηθά να αποκτήσουμε την αλληλεγγύη του σήμερα. Εγώ προσωπικά είμαι περήφανη για το ότι στη χώρα μου, παρά τις έντονες διαβουλεύσεις, καταφέραμε να ξεπεράσουμε το αρχικό σοκ και να κάνουμε έναν πολύ επικοδομητικό διάλογο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ένταξης ε, των μεταναστών. Χρειάζεται λοιπόν αυτό να γίνει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Χρειάζεται να δείξουμε αλληλεγγύη εάν και εφόσον θέλουμε να διατηρήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες μας. Ο κύριος Λόπες Ακυλάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι μεταξύ εκείνων των μελών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που είναι άμεσα και προσωπικά που έχουν κινητοποιηθεί προσωπικά απέναντι σε αυτή την κρίση είναι ανθρωπιστική, αλλά είναι δική μας. Είναι ευρωπαϊκή σε σχέση με την ανταπόκριση, την απάντηση, τη διαχείριση του τι συμβαίνει, του πώς θα διαχειριστούμε αυτό το φαινόμενο, αυτή τη ροή. Και ήταν και το συγκεκριμένο αντικείμενο του δεύτερου πάνελ, δηλαδή η εστίαση του, επί του ρόλου των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων απέναντι σε αυτή την κρίση των αξιών και της ποιότητας της ανταπόκρισης. Οι πολίτες και οι οργανωμένοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν, είναι στην ε, πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Έχουν αναπτυχθεί δίκτυα αλληλεγγύης πολιτών, ακριβώς στην πρώτη γραμμή, εκφράζοντας ακριβώς αυτήν την αλληλεγγύη που κατά τα άλλα ως επίσημο στοιχείο λάμπει δια της απουσίας της. Όμω οι τοπικοί φορείς, οι πόλεις, δεν μπορούν απολύτω τίποτε να κάνουν χωρίς τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών και φορέων. Και πάνω απ' όλα με την απαραίτητη, χρηματοδοτική στήριξη. Όχι μόνο για την δράση πρέπει να λάβουμε στην πρώτη μέρα υποδοχή, αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Βρήκαμε τώρα αυτή τη συμφωνία με τις ποσοστώσεις, λες και αυτό είναι κάποιο είδους λύση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κατανομή ποσοστώσεων με τον ψυχρό τρόπο που το κάνουμε. Προσπαθώ να πω ότι είναι ότι εξακολουθεί να λείπει η δέσμευση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, η κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων, ώστε αυτά τα κεφάλαια της κοινωνικής πολιτικής ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν εγγραφεί στο περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής πρόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υλοποιηθούν. Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα απτά και συγκεκριμένα να εφαρμόσουν ενεγράφησαν 150 εκατομμύρια ευρώ αύξηση στον προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό της κοινωνικής πολιτικής μιλήσαμε και για έναν λεγόμενο μηχανισμό ευελιξίας που θα έδινε απάντηση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τώρα δεν ξέρουμε τι ποσό θα διαθέσει τελικώς η Κομισιόν για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν να στηρίξουν μάλλον τα κράτη-μέλη και τις τοπικούς φορείς και δεν ξέρουμε από πού θα προέρχονται αυτά τα χρήματα. Είναι νέοι πόροι. Από πού προέρχονται, δεν έχουμε απαντήσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι συμμετέχοντες σε αυτήν την διακοινοβουλευτική εδώ συνεδρίαση να έχουμε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή ερωαϊκών αξιών και να είμαστε ικανοί να αναλάβουμε δράση στα εθνικά κοινοβούλια και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προκειμένου να κινητοποιηθούν, να θεσμευτούν αυτοί οι πόροι, να χρησιμοποιηθούν. Και πρέπει να μιλούμε για αξιόπιστα μεγέθη και ρεαλιστικά. Όχι απλώς να αναφέρουμε νούμερα ονομαστικά. Πρέπει να μιλούμε για πόρους λέγοντας από πού προέρχονται, οι οποίοι θα πρέπει να καταλήξουν στο να βοηθήσουν τις συγκεκριμένες προσπάθειες των πολιτών. Ευχαριστώ Χουάν. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξάντλησα τη λίστα των παρεμβενόντων. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια. Ο κύριος Τεκώστερ ίσως θα ήθελε να προσθέσει κάτι στην όλη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι πολλές ερωτήσεις που ετέθησαν είναι ερωτήσεις που δεν απευθύνονται προς την τοπική αυτοδιοίκηση που εκπροσωπώ μέσω της Επιτροπής των Περιφερειών, αλλά απευθύνονται προς τα κράτη και τις εθνικές ε, κυβερνήσεις μας. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί αυτή η αλληλεγγύη. Είναι δυνατότητα, θα έλεγα, αλλά και καθήκον. Καθήκον, επαναλαμβάνω, έναντι της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και που είναι πολύ συχνά αφοπλισμένοι. Καθήκον επίσης και έναντι όσων άκουσα από κάποιους παρεμβαίνοντες και ήθελα να πω ότι θα έβγαινα θλιμμένος από αυτή την ε, ε, συνεδρίαση διότι άκουσα φράσεις που πόρο απήχαν από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να παραμείνουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα στο επίκεντρο. Ευχαριστώ εκείνους που μίλησαν για να καταγγείλουν αυτά που υπόθηκαν, διότι δεν έχουν θέσει αυτά τα λόγια εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, εδώ στο Κοινοβούλιο των Ελευθεριών και πρέπει να πω ότι αυτό ενισχύει ισχύει την ιδέα μου ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και αυτή να προωθήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα και παίρνει τη θέση της με τη γενοδορία που δείχνει. Τα κράτη-μέλη οι κυβερνήσεις που συνεδριάζουν εδώ παράλληλα με τη συνεδρίασή μας και εκεί αυτοί πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Θα πρέπει να ε, μας φροντίσουν να μας ενισχύσουν και να εμποδίσουν εκείνοι που θέλουν να μειγνύουν τα πράγματα. Και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό, διότι ε, αυτοί ε, υπάρχουν και εκείνοι που αντί να θέλουν να λύσουν το πρόβλημα ε, ευημερούν από αυτό και το εκμεταλλεύονται. Η κυρία Κέγκε ίσως θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, όλους τους ε, εισηγητές, όσους πήραν το λόγο και κυρίως το Κοινοβούλιο, τους βουλευτές, τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων που μίλησε στη συνεδρίασή μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στη δουλειά μας με τη συνάδελφό μου τη Ρομπέρτα Ματσόλα για να δεχθούμε όλες τις απόψεις που εκφράστηκαν σήμερα, να τις λάβουμε υπόψη στην έκθεση που συντάσσουμε. Πραγματικά ευχαριστώ από καρδίας και ελπίζω ότι μπορέσουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον τη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ κύριε Κέγκε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου τώρα να πω μερικά λόγια στη μητρική μου ε, γλώσσα, στα βουλγαρικά. Είμαι από τη Βουλγαρία, από μικρή, πολύ μικρή χώρα στην Νότια Ευρώπη. Λοιπόν, είμαι από τη Νότια Ευρώπη και θα να πω ότι σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε στη σημερινή συνεδρίαση. Η χώρα μου και εκείνη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που συνδέονται με την ε, μετανάστευση. Υπάρχουν εκπρόσωποι χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, χωρών που έχουν μακρά παράδοση στον τομέα της ε, μετανάστευσης. Το 2013 η Βουλγαρία εξεπλάγει διότι δεν είχαμε ούτε παράδοση ούτε συνήθεια να ε, εργαζόμαστε με μετανάστες, όμως αποδείξαμε αλληλεγγύη μαζί με όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μια χώρα στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ασφάλεια των συνόρων είναι ασφάλεια, η ασφάλεια των συνόρων μας αφορά την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σήμερα δεχόμαστε επαρκή αριθμό μεταναστών. Εδώ και κάποιους μήνες αυτή την ένθουσα είχα δυνατότητα να πω ότι μετά την τεράστια κρίση της Μεσογείου που δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δεν έχει σταματήσει, πολλοί από τους μετανάστες θα στραφούν, είχα πει, ε, προς τα Βαλκάνια και θα κατευθυνθούν μέσω των Βαλκανίων προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει σήμερα στα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας-Τουρκίας. Ε, δεχτήκαμε τις ε, ποσοστώσεις που διαπραγματεύτηκαν οι ηγέτες χθες. Η Βουλγαρία θα δεχτεί 1.600 άτομα, αλλά μπορώ να σας πω επίσης ότι ήδη δεχόμαστε περίπου 2.000 ε, άτομα την εβδομάδα. Ανήκουμε, συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Ο κύριος Ντεκοστέρ, κύριε Ντεκοστέρ, οι αντιευρωπαϊκές φράσεις που ακούσατε σήμερα δυστυχώς μάλλον ακούστηκαν, αλλά ευτυχώ ανήκουν στη μειοψηφία. Οι περισσότεροι που τοποθετήθηκαν σήμερα, η πλειοψηφία που μίλησαν, οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, καθώ και οι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου, ε, όλοι συμμερίζονται την ίδια προτεραιότητα, απόλυτη προτεραιότητα που είναι η αλληλεγγύη εν ονόματι της ανθρωπότητας και εν ονόματι της Ευρώπης και είμαι σίγουρη ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση και με την βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιμετωπίζουμε πολυάριθμα προβλήματα, αλλά θα καταφέρουμε να τα επιλύσουμε, να πολεμήσουμε μέσω της ενότητας. Σας ευχαριστώ.